Ευχαριστώ πολύ και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία για τις ε, τροπολογίες. Έχουμε δύο τροπολογίες για αιτιολογικές σκέψεις του συναδέλφου Φένιγκεν. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε en Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Και τώρα θα έρθουμε στην τελική ψηφοφορία. Έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όποιος δεν έχει την ε, κάρτα του, παρακαλώ να το δηλώσει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 10 προς 6. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της ψηφοφορίας και θα περάσουμε στο, ε, στο σημείο της ημέρας διάταξη. Υπάρχει μόνο 5 την παρουσίαση τη ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2017. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρόεδρο κύριο Λένε, καλώς ήρθατε, και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Λαζάρου που είναι υπεύθυνο για αυτή την έκθεση και επίσης τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλώς ήρθατε, χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε. Σήμερα είναι ένα σημαντικό, ολοκληρώνει σημαντικό στάδιο. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο, Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Γκρέσλε, κυρία Συγήτρια, αγαπητά μέλη της Επιτροπής, κύριε Πίτροπε, πού βρίσκετε. Ωραία, θα έρθει, θα ήθελα να τον χαιρετήσω. Κυρίες και κύριοι, ως πρώην βουλευτής γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε μια εντατική φάση εργασίας και κάνει προσπάθειες προκειμένου να εκπονήσει διάφορες νομοθετικές πράξεις. Αλλά όχι μόνο αυτό, ε, επίκυνται οι ευρωεκλογέ και είναι το ενδεδειγμένο φόρουμ για το μέλλον της Ευρώπης. Χθες είχαμε, αυτό έγινε σαφέ με τη χθεσινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού τη Εστονία. Εγώ, ω πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που διαθέσετε όσον αφορά τη συζήτησή μα για την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2017. Ο κύριο ε, Λαζάρο, ο οποίο είναι αρμόδιο για την εκπόνηση τη έκθεση και για τα ε, δέκα τη ε, κεφάλαια και Βεβαίω όλα τα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατέβαλαν σημαντικές ε, προσπάθειες προκειμένου να αξιολογήσουμε της, ε, τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού ε, Κοινοβουλίου. Θα παρίσταται εδώ ο κύριος Λαζάρου για τις ειδικότερε ερωτήσεις και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι επεξεργάστηκαν διάφορα κεφάλαια της έκθεσης αυτής. Με αυτή την έκθεση τώρα ξεκινάει η διαδικασία απαλλαγής που είναι η τελευταία κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Ε, θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την συνεργασία τη. Η διαδικασία ελέγχου ε, βασίζεται στην, ε, σε μια αντιθετική διαδικασία παρόλο που δεν είμαστε αντίπαλοι. και ελπίζω ότι ε, εμείς πάντοτε τίναμε δίκον ους ε, στις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, το 2017 καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι αιτήσιοι λογαριασμοί αντανακλούν μια πραγματική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως το προηγούμενο έτος, ε, δίδουμε ένα, μια θετική κρίση όσον αφορά τους ε, αριθμούς ε, για το 2017. Με άλλα λόγια, ένα σημαντικό τμήμα των δαπανών που εξετάσαμε για το 2017 δεν έχει σημαντικό ποσοστό σφαλμάτων. Υπάρχουν δαπάνες για προγράμματα όπου οι δαπάνε χορηγούνται εφόσον πληρούνται ορισμένε προποθέσει. Για παράδειγμα, πληρωμέ για ε, του φοιτητέ του Εράσμου, ε, ε, στήριξη για του γεωργού και μισθή για τους υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι πληρωμές είναι πάνω από το 1,5% του προπολογισμού. Πέρα από αυτό, οι ατασταλίες έχουν μειωθεί το ποστό σφαλμάτων για το 2017 ήταν 2,4% ε, ενώ το 2016 ήταν 3,1% και το 2015 3,8%. Και αυτό καταδεικνύει ότι η οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνει ξεκάθαρα σωστή κατεύθυνση, κάτι που πρωτίστως οφείλεται στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών μελών, επιτρέψατε μου να πω, και στις ε, προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την διεξαγωγή ελέγχων των δραστηριοτήτων του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχω την άποψη ότι, εγώ, ότι εμείς ως ελεγκτές ε, δεν φέρνουμε μόνο κακές ειδήσει, αλλά επισημαίνουμε επίσης υποδειγματικέ διαδικασίες εφόσον υπάρχουν, όπως στην περίπτωση αυτή. Και θα ήθελα ως θετικό παράδειγμα τις άμεσες πληρωμές στο πλάσιο του Ταμείου Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Γεωργία, ε, όπου ε, και για αυτές τις άμεσες πληρωμές ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει κανένα σημαντικό ποσοστό σφαλμάτων. Αλλά στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα επίσης να σε επισημάνω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. Για να σα ξεκαθαρίσω τι εννοώ, θα ήθελα να αναφέρω τρία παραδείγματα. Ένα από ένα άλλο τομέα των γεωρικών δαπανών, το δεύτερο από το τομέα της συνοχής και το τρίτο από το τομέα της έρευνας. Ε, σε μια περίπτωση όπου ένας γεωργός έλαβε μια βοήθεια για τις καλλιέργειες για να καλλιεργήσει τις λεγόμενες ενδιάμεσε ε, καλλιέργειες ωστόσο δεν είχε σωστή λογιστική κάλυψη για το σύστημα άρδευσης κλπ. Και ξεκίνησε μια διαδικασία προκειμένου να ανακληθεί η χορήγηση της ενίσχυσης. Σε μια άλλη περίπτωση ε, κάποιος ε, ευνοούμενος ε, στο πλαίσιο ταμείου συνοχής είχε δηλώσει πολύ, υψηλά, πολύ υψηλές έμεσες δαπάνες πρόκειτο για ε, δαπάνες που δεν ε, τεκμηριώνταν βάσει του ειδικού προγράμματος και δεν είχαν άμεση σχέση με το πρόγραμμα αυτό. Και στην τρίτη περίπτωση μια μικρομεσαία επιχείρηση που συμμετείχε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ε, τις ε, ώρες ε, εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι ώρες εργασίας είχαν ε, μετρηθεί με έναν στρεβλό τρόπο. Έτσι λοιπόν θεωρήθηκαν οι δαπάνες αυτές ως μη χρηματοδοτήσιμες. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι συχνά ε, είχαμε επαρκείς πληροφορίες ε, προκειμένου να εμποδίσουμε ένα μεγάλο σημαντικό ποσοστό των σφαλμάτων και προκειμένου να τα διορθώσουμε. Ενώ οι πληροφορίες που εξοπλίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές, ένα μεγαλύτερο τμήμα ε, του προπολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είχε ένα ποσοστό σφαλμάτων το οποίο ήταν αμεληταίο. Ωστόσο θα πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Τα διοικητικά και ελεγκτικά συστήματα έχουν βελτιωθεί και αυτό μας δίδει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε εκ νέου το πώς ε, οι βελτιώσεις αυτές ε, μπορούν να συμβάλλουν ε, στον, στη διαδικασία ελέγχου. Για το 2017 είχαμε, όσον αφορά την κοινωνική και οικονομική συνοχή, είχαμε μια τροποποιημένη προσέγγιση. σημαντική αλλαγή ήταν ότι οι έλεγχοι οι οποίοι γινόντουσαν στο παρελθόν από τις αρμόδιες αρχές έγιναν εκ νέου αντικείμενο ελέγχου και έγιναν κάποια, έγινε κάποια τροποποίηση στη διαδικασία η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ισχύει για την παρούσα ε, ε, περίοδο. Ε, σε περίπτωση που διαπιστώσαμε κάποιες ατασταλίες, προσπαθήσαμε να τις διορθώσουμε. Έτσι λοιπόν ε, ε, μπορούμε να πούμε βεβαίως να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν ακόμα κάποια ισχνά σημεία τα οποία χρήζουν ε, βελτιώσεων. Τα επόμενα χρόνια θα διευρύνουμε, θα διευρυνθούν θα συμπεριφθούν στον έλεγχό μας και άλλοι τομείς και θα αξιολογήσουμε κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μπορεί να χορηγήσει αυτά αποτελέσματα στους ε, πολίτες της. Ε, δεν αρκεί να πούμε κατά πόσο έχουν δαπανηθεί σωστά τα κονδύλια, αλλά θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουμε κατά πόσο είναι ουσιαστική και έχει νόημα αυτή η απορρόφηση των κονδυλίων ή όχι. Για παράδειγμα, μια, ένας διεθνής οργανισμός έγινε αντικείμενο ελέγχου σε μία τρίτη χώρα και είναι διάφορα παραδείγματα τα οποία δείχνουν ότι είναι δύσκολο να αιτιολογήσουμε στους πολίτες πρόκειται για τα κάποια ε, χρήματα που δαπανήθηκαν για την ε, αξιολόγηση κατά πόσο έγινε σωστά η εκλογική διαδικασία σε μια τρίτη χώρα. Στις ε, περιπτώσεις αυτές είναι δύσκολο να αιτιολογήσουμε στους πολίτες γιατί θα πρέπει τα χρήματα φορολογουμένων να πηγαίνουν σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Για τα προσεχή έτη η Επιτροπή έχει προτείνει μια σειρά από μέτρα που οδηγούν σε μια καλύτερη χρήση των κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής. Ένα τμήμα των ε, προτάσεων θα πάρετε στα σχέρια σας όσον αφορά το πολυθέσιμο συνομικό πλαίσιο. Από την άλλη, εν του ύψου των ε, δαπανών ε, στα οποία έχει δεσμευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται κάτω από έντονε πιέσει Λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το χαμηλό επίπεδο ε, πληρωμών, οι προγνώσεις ε, δείχνουν ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα μπορούσαν ε, οι υποχρεώσεις πληρωμών να αυξηθούν περισσότερο. Ε, η κατάσταση αυτή θα πρέπει να εξεταστεί από μας Στην αντιπαράθεση μεταξύ καθαρών πληρωμών ε, καθαρών πληρωτών συγγνώμη, και καθαρών ε, ε, αποδεκτών, το ελεγκτικό συνέδριο δεν θέλει να αναμειχθεί σε αυτή την αντιπαράθεση. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρχή των οικονομικών προγράμματων, όπου γίνεται αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση μεταξύ των νομοθετών όσον αφορά τις δεσμεύσεις πληρωμών. Αυτό αναβάλλεται στο, για το μέλλον και Προφανώ ε, το αντικείμενο αυτό χάνει την ουσία του. Κυρίε και κύριοι, ε, το σύνολο του προπολογισμού κάνει το 1% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό τα κονδύλια αυτή του ευρωπαϊκού προπολογισμού να χρησιμοποιούνται σωστά. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αξιολογήσουμε ρεαλιστικά τι γίνεται με τα κονδύλια ε, τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Γιατί αν δεν ε, ανταποκριθούμε στις προσδοκίες ε, των ε, πολιτών, θα χάσουμε σε βαθμό αξιοπιστίας. Γι' αυτό θα πρέπει κάθε μέρα να αποδεικνύουμε ότι κάθε αρμοδιότητα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υλοποιείται με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι σε εθνικό επίπεδο. Επιτρέψατε μου να σε αναπτύξω και μία τελική σκέψη πριν ολοκληρώσω την ομιλία μου. Οι ελεγκτέ έχουν την φήμη ότι πάντοτε το βλέμμα του είναι στραμμένο προ το παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι φέτο έχουμε το δικαίωμα να στρέψουμε το ε, βλέμμα μα προ το μέλλον. Στι προσεχεί εβδομάδε θα υπάρξουν γνωμοδοτήσει σε διάφορε προτάσει που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλει για το προσεχέ πολιετές, δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020. Εμείς ε, χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η Επιτροπή εδώ έχει δημιουργήσει μια βάση ε, μεριμνώντας για ένα μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίες, ε, κάτι στοιχείο που απουσιάζει από το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και αυτό είναι σίγουρα ένα βήμα στην ε, ορθή κατεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να ε, φροντίσουμε οι αποφάσεις μας να δράζονται σε μια στέρεη βάση και να δείξουμε στους πολίτες ότι μπορούμε να εκπληρώσουμε τις υποσχέσεις μας και αποτελεσματικά ε, μπορούμε ε, να παράσχουμε απτά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και χαίρομαι για την προσεχή συζήτηση. Είμαι στη διάθεσή σας τόσο εγώ ο κύριος Λαζάρου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε για την πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική σας παρουσίαση. Θα ήθελα να πω ότι παρέλειψα να χαιρετήσω προηγουμένως τον κύριο Έτιγκερ, συγγνώμη, τον κύριο Επίτροπο. Κύριε Λαζάρου, θέλετε να πάρετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος. Ε, Ευχαριστώ όμως να απαντήσω σε ερωτήσει. Ο, Προ... ο Έτιγκερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία ε, Κρέσλε, κύριε Λένε, κύριε Λαζάρου, κύριε Μάρφη, από το ελεγκτικό συνέδριο, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει για την ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και λαμβάνει υπόψη της με μεγάλο ενδιαφέρον τις ε, συστάσεις. Είμαστε ευγνώμονες που το ελεγκτικό συνέδριο ε, πληρεί, ε, ε αποδίδει μια σημασία, συγγνώμη, στον, ε, μεγάλη σημασία στον ρόλο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι το μόνο αλλά ένα καθοριστικό εργαλείο χάραξης της πολιτικής μας και συμμεριζόμαστε το στόχο ε, μέσω των κονδυλίων του προπολογισμού να παραχθεί μια γνήσια ευρωπαϊκή υπεραξία. Τα κονδύλια ε, είναι το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, άρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ε, στοχευμένα και σε στόχους που έχουν, σε αποδέκτες που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά. αυτό δεν είναι εύκολο ε, και δεν είναι εύκολο να το δείξουμε στην κοινή γνώμη. Γι' αυτό είναι σημαντική η μείωση του ποσοστού σφαλμάτων και η, μεγιστο... η βελτιστοποίηση του προπολογισμού με τον τρόπο αυτό. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, το αναγνωρίζει όπως και αναγνωρίζει βεβαίως ότι θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις ή θα μπορούσαν να γίνουν περαιτέρω επιδόσεις. Το 2017 είναι ένα βήμα παραπέρα προς την βελτιστοποίηση της χρήσης των κονδυλίων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Και ανάγεται ε, σε διάφορες συστάσεις του, Ευρωπαϊκού, του ελεγκτικού συνεδρίου από τα περασμένα χρόνια, τα οποία εμείς πράγματι παίρνουμε στα σοβαρά και με τον τρόπο αυτό ε, ε λαμβάνουμε υπόψη μας τις, ε, τις που αναπτύξατε εν σχέση με τι διαδικασίε απαλλαγή τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά τη βελτιστοποίηση τη της των κονδυλίων, υπάρχει μια θετική συνεργασία μεταξύ Επιτροπής και χωρών μελών καθώς και των αρμόδιων αρχιών. Μια τέτοια συνεργασία είναι πολύ καθοριστική και θα βελτιστιοποιήσει περαιτέρω την ε, διαδικασία αυτή, δηλαδή τα αρμόδια μεταξύ αρμοδίων Υπουργείων των χωρών μελών και της ε, Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη. Και εδώ μπορούν να γίνουν βεβαίως ακόμα περισσότερες βελτιώσεις. Γνωρίζουμε τις ε, σκέψεις που διατυπώνονται και τους προβληματισμούς σε σχέση με την ποιότητα και την ορθότητα όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων σε ορισμένε χώρες μέλη. Και το θέμα αυτό επανέρχεται στα τακτά χρονικά διαστήματα ε, στο προσκήνιο, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσπαθούμε να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ε, σφάλματα ή κακή χρήση. Ο κύριος Λένε διαπιστώνει μια εξέλιξη προς την ορθή κατεύθυνση η οποία εκδηλώνεται ως εξής η ελεγκτική διαδικασία του συνεδρίου οδήγησε στο συμπέρασμα μιας μείωσης του ποσοστού σφαλμάτων στα περισσότερα μεγάλα προγράμματα όπου βλέπουμε να υπάρχει μια μείωση του ποσοστού σφαλμάτων. Η συνολική εξολόγηση του ελεγκτικού συνεδρίου ε, ε, όπου για δεύτερη φορά αναγνωρίζεται η βελτίωση στην οικονομική διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική. Μια σειρά βεβαίως παρατηρήσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου δεν είναι νέες, δεν είναι καινούργιες και ε, προσπαθούμε να τις ακολουθήσουμε στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Και μελλοντικά θα έχουμε κατά νου στην περαιτέρω, στο περαιτέρω έργο της ε, Επιτροπής ε, αυτές τις παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, ε, τα δαπάνες του προσωπικού ε, και οι προδιαγραφές είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σωστά. Γι' αυτό θα εξετάσουμε και πάλι τις κατευθυντήριες γραμμές ε, σε συνάρτηση ακριβώς με αυτή την παρατήρηση του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά την πολιτική συνοχή. Εδώ υπάρχουν ελλείμματα όσον αφορά τις αρμόδιες αρχές ε, στις διάφορες χώρες μέλη και μετά από αυτή τη διατύπωση πρόκειται να επικεντρώσουμε το έργο μας στην επαλήθευση της ποιότητας και συμβατότητας του έργου των ελεγκτικών αρχών στο επίπεδο των χαρών, χωρών μελών. Ε, πρόκειται να τα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγυς. Τώρα στο θέμα των ε, δεσμεύσεων των, ε, των ΡΑΛ, των υπολείπων προς εκαθάριση. Εδώ πρόκειται για 270 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ έχω μία ανησυχία. Ε, όσον αφορά το better ε, spending. Ε, ίσως θα μπορούσαν τα χρήματα αυτά να θεωρηθούν ότι είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, αν έρχονται σε όγκο, στο των δύο ετών του προπολογισμού. Η Ευρώπη συνήθως εργάζεται με προγράμματα τα οποία ε, ε, διαρκούν πολλά χρόνια, για παράδειγμα στο πλαίσιο της ε, συνοχής. Μας παρουσιάζονται, τα αξιολογούμε, αναλαμβάνονται δεσμεύσεις, γίνεται προγραμματισμός, εκπονείται το έργο κλπ. Άρα πέντε έτη, τα προβλήματα πέντε έτη δεν είναι υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Και γνωρίζετε για παράδειγμα ότι στη Γερμανία η υλοποίηση προγραμμάτων είναι εξαιρετικά μακρόχρονη γιατί υπάρχουν υπερβολικά πολλές ε, ρυθμίσεις. Ε, το κράτος δικαίου προβλέπει σύνθετες διαδικασίες, γι' αυτό είναι σημαντικό οι υποχρεώσεις να καταλήξουν σε πληρωμές. Ε, αλλά το ποσό αυτό είναι ε, Οι προσπάθειε μα είναι να το μειώσουμε, αλλά δεν είναι κάτι τέτοιο εύκολο, γιατί σας λέω εκ των προτέρων, τελικά ε, το, τα χρήματα αυτά ε, θα είναι λιγότερα. Τα 267 δις είναι μεταβατικός, είναι ένα νούμερο το οποίο δεν είναι οριστικό. Άρα λοιπόν πρόκειται για συνήθεις βραδίες ε, ε, διαδικασίες ολοκλήρωσης ε, προγραμμάτων τα οποία στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ότι σε άλλα κρατικά μορφώματα τα οποία μεν αναγνωρίζουμε αλλά δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι υποδειγματικά. Τώρα, στο επόμενο πλαίσιο του προπολογισμού θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μειώσουμε τη διάσταση αυτή ε, ψηφίζοντας ε, ένα πλαίσιο του προπολογισμού το οποίο δεν θα ισχύσει το οποίο θα ισχύσει τον Απρίλιο του 2019 ενδεχομένως, προκειμένου οι προετοιμασίες όλων των αρμόδιων αρχών να ε, μπορέσουν να ανταπεξέλθουν ε, σε, αυτή το, σε αυτό το χρονικό όριο. Και σας είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας. Αλλά θα ήθελα να σας πω εκ των προτέρων ότι πολλές χώρες μέλη έχουν μια διαφορετική προσέγγιση εδώ και θα ήθελα εν συν 3, εν συν 4 κλπ. Εν συν 2 είναι πιστεύω μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα, όσον αφορά το ποσοστό των σφαλμάτων και την μείωσή του, ε, είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, προσπαθούμε να επιφέρουμε περαιτέρω βελτιώσεις εδώ. Και θέλουμε να τονίσουμε ότι όταν μιλούμε για σφάλματα, δεν πρόκειται πάντοτε για πάτη ή για διασπάθηση ή για διαφθορά. Ε, βεβαίως αυτές είναι οι βαριές περιπτώσεις. Αλλά πρόκειται και για σχεδόν ε, ε, συνήθις, σφάλματα, όχι για περιπτώσεις απάτης. Και ορισμένα ποσοστά σφαλμάτων, ορισμένα ασφαλμένα ποσά ε, δεν αφορούν το, πέρας, το τέλος του έτους, αλλά εμφανίζονται στη διάρκεια του έτους. θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και μετά τη διεξαγωγή όλων των ελέγχων ε, το ποσοστό σφαλμάτων είναι κάτω από το 2%. Το 2017 είναι κάτω από το, εκτιμούμε ότι είναι πάνω από το 1%. Θέλουμε να προσθέσουμε, να προσθέσουμε περαιτέρω τις διατάξεις, αλλά χωρίς να αποδυναμώσουμε τα ελεγκτικά συστήματα. Αυτή είναι η ευκταία ισορροπία. Ή δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία, αλλά αρκετά αυστηρή έλεγχη, ούτε ώστε ε, να μην οδηγηθούμε σε μια αποδυνάμωση του ελέγχου και σε ελλείμματα. Τώρα, όσον αφορά την προσθέμενη αξία, την υπεραξία, ε, ε, εδώ έχουμε κάποιες επιτυχίες και θα μπορούσα, κύριοι βουλευτές, να αναφερθώ για τους ε, ετήσιους ε, για το... σας δείχνω που Ποια είναι τα αποτελέσματα για τον ε, πολίτη. Οι σημαντικές επιτυχίες δείχνουν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, με κάθε ευρώ, με κάθε πρόγραμμα μπορούμε να δημιουργήσουμε μία υπεραξία η οποία ε, δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί μέσω των εθνικών δαπανών. Ε, και θέλουμε να ανταποκριθούμε ακόμα περισσότερο σε αυτό το θέμα του added value, ε, ε, μη προωθώντας κανένα πρόγραμμα το οποίο δεν παράγει τεκμηριωμένα αυτή την προσθέμενη αξία. Και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ε, στο, στη διάσκεψη που θα γίνει, στο συνέδριο που θα γίνει στις 12 Οκτωβρίου θα μιλήσουμε για τις προσπάθειες που θα καταβάλουμε ε, ούτως ώστε να βελτιστιοποιήσουμε αυτή τη ε, διαδικασία. Οι προτάσεις για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο παρέχουν σημαντικές συμβουλές του ελεγκτικού συνεδρίου και της διαδικασίας απαλλαγής Σα είμαι ευγνώμων που το ελεγκτικό συνέδριο δεν στρέφει τη ματιά του μόνο προς το παρελθόν και δεν, αλλά στρέφει τη ματιά του και προς το μέλλον εκπονώντας αναλύσεις εν σχέση με το πώς διαγράφεται το μελλοντικό τοπίο διατυπώνοντας σημαντικές ε, συμβουλές και για το μέλλον ε, όσον αφορά το σχέδιο προπολογισμού για το 2019 ε, και για το ε, και για τη συνέχεια. Βεβαίως η ευελιξία είναι ένας σημαντικός στόχος προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τους καθαρούς πληρωτές ε, και τους καθαρούς αποδέκτες, θέλω τα λεφτά μου πίσω, ε, θεωρώ ότι το αίτημα αυτό δεν είναι πλέον επίκαιρο, γιατί στο παρελθόν η συνοχή και οι γεωρικές δαπάνες ήταν 80% περίπου των δαπανών. Ε, υπήρχαν προγράμματα και ε, ζωφερές πληρωμές αλλά τώρα ε, με, το προσφυγικό, την έρευνα, την προστασία των συνόρων, θέματα τα οποία, των οποίων σημασία αυξάνονται, αυξάνεται συνέχεια, τα χρήματα αυτά δεν ε, έρχονται πίσω, αλλά μένουν στο Μαλί, στα σύνορα Τουρκίας, Βουλγαρίας κλπ. κλπ. Αλλά με τον τρόπο αυτό εκπληρώνουν οι προσδοκίες των χωρών μελών και των πολιτών χωρίς να επιστρέφουν στα ταμεία των χωρών ε, μελών. Ε, και με τον τρόπο αυτό ε, οι φορολογούμενοι ε, στις χώρες πληρωτές γνωρίζουν ότι τα χρήματα αυτά πηγαίνουν στην, στους σωστούς, στους κατάλληλους αποδέκτες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να ολοκληρώσω λέγοντας ότι την επόμενη εβδομάδα θα εξετάσουμε κατά πόσο η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου μπορεί πραγματικά να συμπεριληφθεί στην βάση του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βλέπω να υπάρχουν εδώ καθόλου εμπόδια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ε, θα, θα, θα, να κάνουμε τώρα έναν γύρο των εισηγητών και μετά των σχεδόν και στη συνέχεια όλα τα μέλη της Επιτροπής. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Ιάλα Σάντερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Λένε και τον κύριο Λάσαρο για αυτή την ε, ετήσια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου που παγιώνει μία τάση που είχε ήδη διαμορφωθεί στο παρελθόν μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων Ελεγκτικού Συνεδρίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ε, έδωσε μεγάλη μάχη μπροστά στις επικρίσεις και συστάσεις και θα πρέπει να σκεφτούμε και τα κράτη-μέλη τα οποία κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθούν σε αυτό το έργο όπως μας είπε και ο Επίτροπος Έτιγκερ. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχει επιτελεστεί πρόοδος και φυσικά πολλοί ψεύδονται ως προς την κατάσταση και τον τρόπο εφαρμογής ενός προϋπολογισμού που αφορά το 1% όπως είπε και ο κύριος Λένε, το 1% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο και μελλοντικά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύουμε ήδη το δέκατο έτος της. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε πώς ε, μπορεί να εφαρμοστεί ένα δημοσιονομικό πλαίσιο με βάση ε, μία θετική έκβαση εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτική, γιατί σίγουρα παγιώνεται μία στάση λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 ο όγκος πληρωμών μειώθηκε, αλλά από την άλλη πλευρά είδαμε ότι έγινε πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων. Εξακολουθούμε να ζητούμε από το ελεκτικό συνέδριο να ε, συνεχίσει με αυτή την θετική τάση και θεώρηση του ζητήματος. Είναι γεγονός ότι η δική μας Επιτροπή ζήτησε πληθώρα μεταρρυθμίσεων από το ελεγκτικό συνέδριο και το ελεγκτικό ε, αναθεώρησε τις δραστηριότητες του σε θέματα που αφορούν την ευημερία των πολιτών. Παρ' όλα αυτά όμως αντιμετωπίζουμε ορισμένες δυσκολίες γιατί ως προς την ΚΑΠ και την συνοχή θα πρέπει να συνεργαστούμε έτσι ώστε να βασιστούμε στα αμοιβαία στοιχεία που χορηγούμε μεν στους δε. Και φυσικά να καταπολεμήσουμε και αυτή τη στάση των ευρωφοβικών και ευρωσκεπτικιστών. Νομίζω ότι αυτή αυτό είναι μέρος της εργασίας για την απαλλαγή. Φυσικά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις άμεσες πληρωμές ή τις αποζημιώσεις και επιστροφές στα πλαίσια του, του περιθωρίου αυτού σφάλματος. Και φυσικά μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξαναδούμε τις επιστροφές ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει θέμα διαχείρισης. Πρέπει να βελτιώσουμε το διαχειριστικό αυτό πλαίσιο και όπως έχουμε πει εδώ και χρόνια, θα πρέπει να διεξαχθούν επιτόπιες έρευνες ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινή διαχείριση. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πάντα βέβαια, γιατί στη δημοσιονομική διαχείριση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ταχύτητα διαχείρισης της ε, κρίσης και φυσικά τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, τα ραλ, έχουν ε, αυξηθεί ουσιαστικά. Γι' αυτό θα πρέπει και στα πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κοινή διαχείριση για να μην ε, επιπέσουμε στα ίδια σφάλματα που είναι δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες. Στο θέμα της ε, συνοχής αντιμετωπίζουμε θέματα προθεσμιών. Και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική έλλειψη διαφάνειας στον προϋπολογισμό. Θα πρέπει να συνεργαστούμε εκ του σύνεγγυς ε, με το ελεγκτικό συνέδριο, εκεί που δεν υπάρχει κοινό έδαφος συνεννόησης. θα πρέπει να ε, διαχειριστούμε και το θέμα του μεταναστευτικού. Μέσα στα πλαίσια και της ανάπτυξης, διότι η μετανάστευση έχει και εσωτερικό και εξωτερικό άξονα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εμείς ε, όταν σταθμίζουμε τα πράγματα θα πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα αυτό τον προϋπολογισμό για τη μετανάστευση, ο οποίος είναι ιδιαίτερα περιορισμένος, όμως τα συνοδευτικά μέτρα δεν βοήθησαν ιδιαίτερα ώστε οι πολίτες να κατανοήσουν την προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού για να εξευρεθεί μία σωστή λύση για το μεταναστευτικό. Θα πρέπει να εξηγήσουμε στους πολίτες πώς διαχειριζόμαστε αυτό το θέμα. Το 2019 θα προκύψει μία νέα συζήτηση αναγνώρισης επιμέρους προβλημάτων, αλλά φυσικά ο λαϊκισμός πολλές φορές επικρατεί. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε, να επεξηγήσουμε πώς αυτός ο προϋπολογισμός και αυτές οι δράσεις αποτελούν ένα ε, στοιχείο μόχλευσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ζητήματα και μετά τις εκλογές. Αυτό είναι το θέμα το οποίο τονίζουν οι λαϊκιστές, βασίζονται σε αυτό. Γι' αυτό νομίζω ότι στα πλαίσια της απαλλαγής θα πρέπει να δούμε τι ορίζοντα θα δώσουμε σε αυτές τις άλλες ε, δραστηριότητες, το νομοθετικό σκέλος, την ΚΑΠ και την ε, διαχείριση. Πρόκειται για μοχλούς που θα μας βοηθήσουν για να διαχειριστούμε αυτό το 1% του προϋπολογισμού και το οποίο έχει πολλαπλές συνέπειες. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Λέινε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γιάλα. Θα ήθελα να πω μόνο ε, κάποιες παρατηρήσεις, τέσσερις παρατηρήσεις συμπληρωματικά. Το ένα, είναι τεράστια πρόοδος όταν η Επιτροπή προτείνει σε σχέση με τα υπόλοιπα προς εκαθάριση μεταβαίνουμε από το 1 συν 1 στο 1 συν 2. Το 1 συν 3 η διαδικασία έγινε γιατί μετά την κρίση πολλές χώρες μέλη είχαν ε, τεράστια προβλήματα όσον αφορά τα επιπρόσθετα κονδύλια. Γι' αυτό θα πρέπει να, φύγουμε από αυτή την περίοδο που έγιναν κάποιες εξαιρέσεις. Τα ραλ, τα υπόλοιπα προς εκαθάριση ε, υπάρχουν σε κάθε προϋπολογισμό. Ε, τώρα πλέον είμαστε σε μια κατάσταση όπου το ποσό αυτό είναι το διπλό του προϋπολογισμού και βεβαίως αυτό δημιουργεί κάποιες αβεβαιότητες. Ε, δεν είναι ιδεώδης η κατάσταση. Εξού και παράκληση και ε, να αναστραφεί η τάση αυτή και ελπίζω ο νομοθέτης να ακολουθήσει και μπορώ να φανταστώ ότι ορισμένες ε, χώρες θα ήθελαν εν, νη, συν, αλλά δεν γίνεται. Η διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει θεωρώ λοιπόν ότι είναι σωστή αλλά θα πρέπει πράγματι να εφαρμοστεί σωστά. Και θα ήθελα να σε επισημάνω ότι βεβαίως ε, ε, υπάρχουν δύο τάσεις από τη μία πλούστευση από τη μία μέσω άμεσων πληρωμών από την άλλη το ζήτημα της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεων. Και εδώ θα πρέπει να επιτευχθεί μια ισορροπία. Δεν είναι πάντοτε σωστό να γίνει απλούστευση. Ε, η δασκέρχη ισχύει, αλλά δεν γίνεται πάντοτε. Και προκειμένου ορισμένε φορέ, για παράδειγμα, να γίνουν αποτελεσματικοί έλεγχοι, θα πρέπει να υπάρχει και ένα επίπεδο περιπλοκότητας. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι τόσο ε, υψηλό ο βαθμό, αυτό ο βαθμό περιπλοκότητα, ούτω ώστε να διαπράττονται σφάλματα. Εδώ θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά τη διαδικασία απαλλαγή. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας ε, θα σας υποστηρίξουμε όσον αφορά δε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, όπως είπα την περασμένη εβδομάδα, θα υπάρχει μια σειρά γνωμοδοτήσεων από τη δική μας πλευρά. Ελπίζω να τις αξιοποιήσετε σωστά. Και το θέμα των υπολείπων προς καθάριση θα υποβληθεί επίσης σε μια προσεκτική ανάλυση εγώ ως πρόεδρος του ελεγκτικού συνεδρίου θα πω στους συναδέλφους να δούμε κατά πόσο δεν θα έπρεπε να προβούμε σε μία ανάλυση των λόγων για το οποίο είναι τόσο υψηλό το ποσό των υπολείπων προς εκαθάριση και να διατυπώσουμε κάποιους προβληματισμούς εν σχέση με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση αυτή. Για παράδειγμα, η έκθεση για το Jaspers, ένα εργαλείο το οποίο είχε σαν σκοπό να βελτιώσει τις διοικητικές ικανότητες των χωρών, ικανότητα, την ικανότητα των χωρών μελών να προβούν σε μια καλύτερη διαχείριση προς επίτευξη αυτού του στόχου. Το θέμα της μετανάστευσης βεβαίως ε, είναι ένα μια νέα προτεραιότητα. Το τρίτο σώμα πλέον δεν ε, εξετάζει μόνο θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και κράτου δικαίου, μετανάστευσης και άλλα θέματα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια... είναι υπεξεργασία με έκθεση για το ζήτημα της μετανάστευσης, το οποίο... η οποία θα ολοκληρωθεί ε, σύντομα και η οποία θα επαβάλει συγκεκριμένε ε, προτάσεις βελτίωσης από την πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ. Τώρα θα έρθουμε στο γύρο των σκιωδών. Επειδή εγώ είμαι σκιώδης του ΕΛΚ, θα πάρω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Είναι μια χρήσιμη έκθεση, αλλά φράσεις επαναλαμβάνονται σε όλες τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Ότι η Επιτροπή δεν αξιοποιεί τις πληροφορίες που έχει, επαρκώς τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Ε, έχει διατυπώσει κάποια απόθεση εργασία στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με αυτό το φαινόμενο. Γιατί δεν αξιοποιεί η Επιτροπή τι ε, πληροφορίε αυτέ. Κύριε Επίτροπε, γιατί δεν αξιοποίησατε τις ε, ερωτήσεις, τα στοιχεία, που, τις πληροφορίες που είχατε στη διάθεσή σας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα και σχέση με το πώ θα μπορούσε να περάσει αυτό τι χώρε μέλη. Δεύτερον, οι ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις όσον αφορά την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Το θέμα τη αξιοπιστίας των στατιστικών στοιχείων. Και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες προ την Κομισιόν, η οποία έχει αναγνωρίσει εδώ και πολύ καιρό το ζήτημα αυτό. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά ως προς την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων και της κριτικής που κάνατε στην ενετήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Τρίτον, τα οικονομικά εργαλεία. Νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον ζήτημα. Ε, οι δαπάνες εδώ έχουν τετραπλασιαστεί, αλλά τα κονδύλια τα οποία τελικά φτάνουν στα χέρια των ενδιαφορεόμενων είναι κάτω από 10% υπάρχει εδώ ένα νομικό χάσμα. Γιατί τα χρήματα δεν αρκούν. Έχουμε μόνο παλαιούς αριθμούς, πολύ παλιές εκθέσεις με στοιχεία. Ποια είναι λοιπόν τα δικά σας συμπεράσματα εδώ για τα οικονομικά εργαλεία, γιατί θεωρώ ότι είναι λυπηρό, λυπηρή η κατάσταση γιατί πρόκειται εδώ για έναν γρήγορο τρόπο διεξαγωγής των επενδύσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο και τελικά στην πραγματικότητα γίνεται το αντίθετο. Και εμείς εδώ πάντοτε το ζούμε σαν φιάλτη. Πέντε είναι, ας πούμε, υπάρχει ένα ποσό πέντε δις για που δεν ξέρουμε τι έχει απογίνει. Άρα λοιπόν τι θα έπρεπε να κάνουμε κατά την άποψή σας. Τώρα, για την έρευνα το ποσοστό σφαλμάτων είναι υψηλό 4,2%. Ποια είναι εδώ τα συμπεράσματά σας. Θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι είναι απελευθερωτικό αυτό που μας είπατε, ότι συνολικά μειώνεται το ποσοστό των ε, σφαλμάτων. Ε, θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό αυτό. Ε, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συν. Αλλά διαπιστώνουμε ποιος είναι ο τεράστιος ρόλος των προχρηματοδοτήσεων. Ε, και ίσως ε, θα πρέπει να το δούμε αυτό. Από το Άλντε τώρα είναι η Μαρτίνα Λεμπαγιώβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε να ευχαριστήσω πρώτον το Ελληνικό Συνέδριο για, την, για το εξαιρετικό έργο τους με τη μορφή της έκθεσης του 17. Για μένα, όπως θα περιμένετε, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία που αφορούν την απόδοση και τις επιδόσεις. Για, για την άλλη, εδώ και χρόνια είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Το σχετικό κεφάλαιο αποτελεί για μας προσθέμενη αξία. Η Κομισιόν δυστυχώ δεν χρησιμοποιεί, δεν αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες εγκαίρως και λυπούμε για το ότι η Κομισιόν δεν είναι αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να δρομολογήσει τις απαραίτητες διορθωρικές δράσεις. Η Κομισιόν θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα. Και αυτό λέω και εγώ εδώ σήμερα. Πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα, εσωτερικά και εξωτερικά, με γνώμονα τις υψηλότερες δυνατές επιδόσεις. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία και για την Κομισιόν. Και αυτό το οποίο με εξέπληξε επίση στην έκθεση είναι το γεγονό: ότι η δομή των δαπανών παραμένει η ίδια. Δηλαδή όλα τα σφάλματα όσον αφορά τις ανακτήσεις ή τα μη επιλέξιμα προγράμματα ε, αφορούν τις ίδιες κατηγορίες, 93%. Παρά τις ε, προσπαθείς απλούστευσης, θέλω να πω ότι αν οι αρχές μας δεν μπορούν να επιλέξουν μεταξύ επιλέξιμων και μη έργων, προφανώς θα είναι δύσκολο για τους ε, δικαιούχους. Οπότε το πρώτο ερώτημά μου βαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση, τη δομή του σφάλματος, το περιεχόμενο του σφάλματος και ρωτώ το ελληνικό συνέδριο, τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε το βαθμό κατανόηση, να καταλαβαίνει ο κόσμο τι είναι επιλέξιμο έργο, τι είναι επιλέξιμη δαπάνη. Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα μπορέσουμε, πιστεύω, να αποφύγουμε το 90% των σφαλμάτων στην χορήγηση ενισχύσεων. Και επίσης, δεύτερον, έσοδα. Θα ψηφίσουμε απόψε για θέματα τελειωνιακά, εσόδων, απάτη κλπ. Είναι τα θέματα τα οποία παρέρχονται κατά κόρον στο ελληνικό συνέδριο, στα τη Όλαφ, στι εκθέσει του κλπ. Ερωτώ το συνέδριο, το ελληνικό συνέδριο, πώς θα συλλέξουμε σωστά, πώς θα εισπράξουμε σωστά ε, τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους της Ένωσης, σε όλα τα σημεία στα οποία εισπράττουν αυτή, τη Φλάναγκαν, Δε Γιόγκ μετά. Κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη, ο αδερφός μου έπρεπε να φύγει. Θα με βάλουν σύντομο. Η γενική εικόνα είναι θετική. Νομίζω όλοι συμφωνούμε με αυτό. Καταγράψαμε τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Έχω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά το Ταμείο Συνοχής. Τα κονδύλια του Ταμείου συνοχής. Πέρσι υπήρχε μια υποσημείωση, θα τη βρούμε, που έλεγε ότι στο σφάλμα δεν έχουν συμπολογιστεί οι εκταμιεύσεις προς διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, 2,5 δισεκατομμύρια παρακαλώ, που ήταν τελικώς εκτός περίοδου επιλεξιμότητας σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου. Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσό φέτος γιατί το συζήτησαμε εκτενώς στην Επιτροπή μας. Πού θα πάνε, πού θα προσθεθούν αυτά τα κονδύλια, δεν είναι νόμιμα, δεν είναι επιλέξιμα. Και αυτό θα μας πήγαινε σε ένα ποσοστό σφάλματος 2%. 2% επιπλέον του ποσοστού σφάλματος που έχει καταγράψει, που έχει μετρήσει το ελεκτικό συνέδριο. Επίσης, παρατήρησα ότι στον τομέα ασφάλεια και ηθαγένεια το θέμα δεν περιλαμβάνεται θα σας καλούσα να αλλάξει αυτό του χρόνου. Πρόκειται για έναν τομέα υψηλή σημασία εν ώψη Το συζήτησαμε με την υπηρεσία Σύλλου και εν ώψη μελλοντικών εξελίξεων, διότι όλο και περισσότερα κονδύλια θα δαπανώνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ο τομέα πρέπει να τύχει υψηλότερη προτεραιότητα από τη φέτο. Και τρίτον, ε, για το Ταμείο το λεγόμενο Ταμείο Juncker ανησυχώ. Δεν βλέπω πληρωμές. Συζήτησαμε για τον Benelux βεβαίω, εκεί βλέπω στοιχεία. Αλλά εκεί που χρειάζεται να πάνε τα λεφτά, δεν βλέπω. Ε, βλέπω να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση, μεγάλη ιστέρηση. Μήπως αυτό σημαίνει τελικά στην πράξη ότι το ταμείο αυτό δεν λειτουργεί, δεν αποδίδει. Μήπως θα έπρεπε να θέσουμε υπό αμφισβήτηση την ίδια τη δομή αυτού του ταμείου. Τι μπορούμε να βελτιώσουμε προκειμένου. Ευχαριστώ. Collega Staes, bitte. Dank u, voorzitter. Eerst en vooral wil ik de heer Lene en al zijn aanwezige collega's bedanken voor het goede werk. Niet alleen jullie zelf. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λένε και όλους τους συνεργάτες του. Πολλές φορές ξεχνάμε ότι ότι πίσω από κάθε μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου υπάρχει προσωπικό το οποίο συνδράμει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και χαίρομαι και για την πρότασή σας για τους οργανισμούς ένα μήνα νωρίτερα από ότι πέρσι. Τώρα, ως προς την έκθεση καθεαυτή, τη διαβάσαμε και τα πράγματα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μείωση του ποσοστού σφάλματος κάθε χρόνο, όλο και περισσότερο, όμως υπάρχουν πολλές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες που γνωρίζουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά που δεν χρησιμοποιούνται για τη μείωση του περιθωρίου σφάλματος. Αν δούμε τα στοιχεία για, ε, για, το, σφάλ, για το ποστό σφάλματος για την ανάπτυξη που είναι 4,6% και 2% αντιστοίχως για την ανάπτυξη και την έρευνα, θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα χαμηλότερα ποσοστά όμως ε, πρόκειται για έναν προϋπολογισμό 4 δις. Τώρα το ελεγκτικό μας λέει ότι το ποσοστό σφάλματος είναι 4,5%. Αν όμως είχαν ληφθεί υπόψη αυτές οι πληροφορίες θα είχε μειωθεί στο 2,8%. Όπως είπε η κυρία Γκρέσλε θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε οι κρατικές αρχές να χρησιμοποιήσουν υποχρεωτικά τις διαθέσιμες πληροφορίες γιατί προτείνονται διάφορες μέθοδοι αλλά δεν συμφωνούν τα κράτη-μέλη. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ είχε απόλυτο δίκιο θα πρέπει στην ε, έκθεσή μας να προτείνουμε μία συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να μας απασχολήσει είναι η περαιτέρω αύξηση των ε, υπολείπων ε, προς εκαθάριση, των ΡΑΛ, σελίδες 16 και 17 του εγγράφου που λάβαμε χτες. βλέπουμε ότι υπάρχει ένα υψηλότερο ποσοστό στο τέλος του πολιετούς. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι πιστώσεις υποχρεώσεων δεν θα χρησιμοποιηθούν πλήρως. Μιλάμε για 270 δις. Και αν δούμε τους πίνακες όπου έχετε μια σειρά κρατών και συγκριτικά στοιχεία βλέπω ότι ένα 10% ε, υποπίπτει σε υψηλότερο σφάλμα. Πρόκειται για τις νέες χώρες, άρα το θέμα είναι και πολιτικό, γιατί θα πρέπει να γίνει μία συζήτηση και στα πλαίσια του πολιετούς, έτσι ώστε να γνωρίζουμε πολύ καλά πού και πώς μεταβαίνουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα έχει πολιτική χρειά, ιδιαίτερα για μια σειρά κρατών. Ορισμένες χώρες, λοιπόν οι νέες χώρες, ακόμα δεν χρησιμοποιούν τη σωστή μεθοδολογία. Και υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν υπάρχει στην έκθεση. Κύριε Λένε, θα ήθελα να μου πείτε ποιο είναι, τι γίνεται με το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου ε, για το οποίο γίνεται έρευνα από την Όλαφ. Αυτό απασχολεί τον κόσμο ιδιαίτερα. Πώς προχωρά αυτή η έρευνα. Έχουν υπάρξει πολύ σοβαρές κατηγορίες κατά αυτού του μέλους και μέσα στα πλαίσια της 12ετούς ε, ε, φοιτείας δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μεμονωμένο το επεισόδιο. Νομίζω ότι στο παρελθόν υπήρχαν και άλλα τέτοια κρούσματα. Ελπίζω να έχετε λάβει μέτρα αντιμετώπισης, αλλά δυστυχώς υπήρχε μια τέτοια συλλογιστική στο ελεγκτικό συνέδριο που κατέστησε δυνατή αυτή την κατάχρηση. Δηλαδή δεν πρέπει να βρούμε τον αποδίοπομπαίο και μόνο. Ο Γενικός Γραμματέας επίσης ε, είναι υπεύθυνο αν δεν γίνονται επαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι. Πώς έγινε κάτι τέτοιο για 12 συναπτά έτη. Αυτό σας ρωτώ λοιπόν και θα ρωτήσω και την όλα αυτήν ίδια. Θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, άλλα τέτοια κρούσματα και θα ήθελα η Όλαφ να διερευνήσει όλα τα μέλη εκείνο το χρονικό διάστημα για να δούμε κατά πόσο αυτή ήταν μια κοινή πρακτική και δεν αφορούσε ένα και μόνο μέλος. Πρόεδρε, Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Θα πρότεινα ο κύριος Λαζάρου να πάρει θέση στα ειδικά ερωτήματα και εγώ να συμπληρώσω αν δεν έχουν καλυφθεί όλα. Για παράδειγμα, στην τελευταία παρέμβαση να πω κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, να απαντήσω πρώτα τα ερωτήματα της κυρίας Γκρέσλα και του κυρίου Στάς βεβαίως. Για ποιο λόγο η Κομισιόν, ενώ έχει στα χέρια της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, δεν διορθώνει σφάλματα. Δεν αφορά μόνο αυτό, ξέρετε, την Κομισιόν, αλλά και τις αρχές των κρατών μελών. Γι' αυτό και δεν υπάρχει μία ενιαία απάντηση γιατί τούτο συμβαίνει. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί πει η εσφάλματα καταγραφή των στοιχείων, έλλειψη σαφών οδηγιών από την Κομισιόν, ανεπαρκής εκπαίδευση των στελεχών των ελεγκτικών αρχών σε επίπεδο κράτου μέλους, ανεπαρκής ενδεχομένως εποπτεία από πλευράς Κομισιόν των αρχών των κρατών μελών. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα από το τρέχον έτος σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα μέσω χρηματοδοτικού μηχανισμού που αφορούσε την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βρήκαμε ότι 80% του ποσού ε, πήγε σε επιχειρήσεις που δεν ήταν μικρές. Οι ελεγκτικές αρχές βεβαίωσαν ότι τα χρήματα είχαν αποδοθεί στον χρηματοδοτικό μηχανισμό, αλλά δεν έκαναν τίποτα για, το, για το περαιτέρω. Όταν η Κομισιόν λοιπόν πήρε στα χέρια της την ε, δέσμη των εγγράφων για την ετήσια καθάριση από τα κρατημέλη, δεν επιβεβαίωσαν αυτήν την πληροφορία. Ε, απλώς την παρέλαβαν. Το οποίο σημαίνει ότι εάν είχαν κάνει επιπλέον προσπάθεια, το ποσοστό σφάλματος θα ήταν πολύ χαμηλότερο από το σημερινό. Κύριε Ραπαγεύα, αναφερθήκατε στο τι μπορεί να γίνει για να μειωθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος που προκύπτει από μη επιλέξιμα έργα και μη επιλέξιμες δαπάνες. Η απάντηση είναι και εδώ ίδια περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη υποπτία από την Κομισιόν. Κύριε Κλαπαγιώβα, επίσης ρώτησε τι μπορεί να γίνει ώστε οι δεσμοί να εισπράττονται με τον σωστό τρόπο. Η Κομισιόν πρέπει να φροντίσει ότι υπάρχουν υπαρκείς δυνατότητες διαθέσιμες έτσι ώστε οι τελωνιακοί δεσμοί να εισπράττονται στο σωστό επίπεδο. Και κύριε Ντεγιόγκ, αναφερθήκατε στο ζήτημα που τονίσαμε και πέρσι στην εκθέσή μας σχετικά με τα περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί στον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος λόγω της μετακίνησης της ημερομηνίας εντός της οποίας έπρεπε, πριν από την οποία έπρεπε να αξιοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Αυτό έγινε μία φορά σε διάπαξ, η παράταση δηλαδή της περίοδου. Ε, γι' αυτό και φέτος ευτυχώς δεν έχουμε, δεν αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση. Ο κ. Δεγιόν επίσης αναφέρθηκε σε ένα άλλο θέμα. Την αξιολόγηση του τομέα να αξιοποίηση, αν θέλετε, του τομέα ασφάλεια ηθαγένεια. Έχουμε περιορισμένους πόρους, εν προκειμένου. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε με αυτά τα περιορισμένα κονδύλια. Οι δαπάνε του τομέα είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια. Πιστεύουμε ότι δεν θα προσφέρουμε κάτι αν κάναμε αυτή την αξιολόγηση σε αυτή τη φάση. Όμως, συλλέγουμε τα στοιχεία τα οποία ζητήσαμε για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνολικότερη αξιολόγηση. Όπως, όπως όμως είπε και ο Πρόεδρος, έχουμε διενεργήσει ελέγχους επίδοσης και σε αυτόν τον τομέα και όπως εξήγησε και ο Πρόεδρος, η εντολή του τρίτου τμήματος για να ασχοληθεί ακριβώς και με αυτά τα θέματα. Ο κ. αναφέρθηκε επίση. μάλλον έθεσε ένα ερώτημα αν θέλετε, περί του Ταμείου Juncker. Αν δηλαδή το Ταμείο Juncker κάνει τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκε. Πολύ σύντομα, πριν από τα τέλη του έτους, θα δημοσιεύσουμε ειδική έκθεση, έκθεση επίδοση σχετικά με το Ταμείο Juncker, όπου θα δηλώνουμε που πηγαίνει το Ταμείο και πώς έχει αποδώσει ως τώρα, αν έχει πετύχει δηλαδή τους στόχους του. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λάζαρου. Νομίζω έχουν μείνει κάποια σημεία ανοιχτά, τα οικονομικά εργαλεία. Ε, σύντομα θα ε, κατατεθεί, θα παρουσιαστεί η έκθεση εν σχέση με το πόσο αποτελεσματικά είναι τα οικονομικά εργαλεία, ε, πώς γίνεται η κατανομή κλπ. Θεωρώ ότι θα δοθούν συγκεκριμένες ε, απαντήσεις στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή στοιχεία από τη δική μου άποψη, δική μου οπτική γωνία, αλλά θα ήθελα ε, να το συζητήσω συγκεκριμένα ε, όταν ε, υπάρχουν ακριβή στοιχεία, ακριβή νούμερα. Όσον αφορά την, τις επιδόσεις, την, την αποτελεσματικότητα της αιτήσεις έκθεσης, είναι αρκετά καλή, αλλά θέλουμε να κάνουμε περισσότερες βελτιώσεις και θα έχουμε μια συζήτηση σχέση με μια συγκεκριμένη πρόταση ενός συναδέλφου για το πώς η έκθεση αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχουν πολλές ιδέες ε, οι οποίες πρόκειται να συζητηθούν ε, και ε, νομίζω ότι το στηρόχρονο διάγραμμα που έχουμε μπροστά μας μπορεί να εκπληρωθεί και μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνει. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε σε ποια κατεύθυνση θα πάει η συζήτηση. Πάντως θα γίνει συζήτηση πώς μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η, να βελτιωθούν οι επιδόσεις αυτών των, ε, αυτής της έκθεσης. Τώρα, όσον αφορά την μετανάστευση, θα πρέπει σίγουρα να δούμε ε, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε εδώ την ε, διαχείριση. Βεβαίως συνιστά μια προτεραιότητα. Το τρίτο μας σώμα ε, έχει το θέμα αυτό στο επίκεντρο του έργου του και θα έχουμε τα προσεχή χρόνια ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Γιατί όπως είπε ο κ. Ντεγιόγκ, είναι μείζονος ε, πολιτικής σημασίας το ζήτημα και βεβαίως ε, χρειάζεται να ασχοληθούμε και θα παρακολουθήσουμε την ροή των χρημάτων ε, καθ' όλη την πορεία της, ούτως ώστε να αξιολογήσουμε το ζήτημα της αποτελεσματικής χρήσης. Τώρα, ε, για το τελευταίο θέμα μπορώ να πω μόνο μια, να κάνω μια παράτηση γενικής φέσεως. Το ζήτημα αυτό λαμβάνεται πολύ σοβαρά. Εξετάζουμε τα πράγματα και θα ε, καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και πρόκειται να εκπονήσουμε μια έκθεση την οποία προτίθεμαι να σας παρουσιάσω. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω περισσότερα πράγματα ως προς οι λεπτομέρειες, γιατί βρισκόμαστε σε μια δημόσια συνεδρίαση εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα... Για την Όλαφ ήταν η τελευταία παρέμβαση. Οι συντονιστές θα ασχοληθούν με το θέμα αυτό, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, ε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα δώσω μία σύντομη απάντηση από τη δική μας ε, πλευράς. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, ε, εκεί το περιθώριο σφαλμάτων ανέβηκε από το 3,3 στο 4,5. Αυτό το, λαμβάνουμε το παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Αλλά βεβαίως εδώ τα προγράμματα έχουν υλοποιηθεί με κάποιους εταίρους οι οποίοι έχουν, τείνουν να αναλαμβάνουν υψηλούς κινδύνους. Πρόκειται επίσης για πολύ, πολύπλοκα προγράμματα και όπου η εμπειρία βελτιώνεται κατά την εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων. Γι' αυτό είναι σημαντικό μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ε, και εφόσον απαιτηθεί η επιστροφή χρημάτων να διατυπώσουμε η οριστική, το οριστικό ποσοστό σφαλμάτων το τελευταίο χρόνο ήταν 1,8. Άρα ε, αποδεκτό. Δεύτερον, κατά πώς αξιοποιούμε όλες τις πληροφορίες. Ε, θα έλεγα εν συντομία ναι. Ε, πραγματικά τις διαβάζουμε, τις ακούμε και τις λαμβάνουμε υπόψη μας. όταν ε, ε, παίρνουμε πληροφορίες για το 2017 δεν ε, μπορούν να αξιοποιηθούν με ορατό τρόπο ήδη μέσα στο 2017 γιατί χρειάζονται μια επεξεργασία. Οι υπηρεσίες μας είναι, δουλεύουν πολύ αξιόπιστα αλλά χρειάζονται ένα περιθώριο χρόνου. Δεν μπορεί να είναι τόσο ταχύ ο χρόνος επεξεργασία. γιατί θέλουμε να καταλήξουμε σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά εργαλεία σε εθνικό επίπεδο, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, γιατί δεν έχουμε μόνο το ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και το εθνικό και το περιφερειακό, που τρέχουν σε τέτοια καινοτόμα οικονομικά εργαλεία. Με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προτείναμε ε, η πρόσβαση σε ελεκτικές ε, δυνατότητες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να διευρυνθεί και σε εθνικό επίπεδο όσο το θέμα της υποχρεωτικής εκπόνησης εκθέσεων για τις χώρες μέλη θα ενισχυθεί στο προσοχές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και παρακαλώ μας υποστηρίξετε ούτε ώστε αυτή η διεύρυνση της υποχρεωτικής εκπόνησης εκθέσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να υποστηριχθεί από τη δική σας πλευρά και να μην αποδυναμωθεί. Ε, ε, όταν πρέπει να ε, είναι ευρωπαϊκό το συμφέρον να γίνεται σωστά η ίσπραξη, να, γίνει, να λειτουργούν σωστά συγγνώμη, τα, οι τελωνιακές υπηρεσίες. Αλλά όσον αφορά την ε, προσπάθεια, τη διαδικασία εξοικονόμησης, ε, ε, στο πλαίσιο μάλλον, συγγνώμη, της διαδικασίας εξοικονόμησης, τελικά οι τελωνιακές ε, υπηρεσίες έχουν ε, ε, συρρυκνωθεί, έχουν περιοριστεί. Άρα εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους και θα πρέπει να ελέγξουμε αποτελεσματικά πώς μπορούμε να εξυπηρετήσουμε το ενδιαφέρον των χωρών για να έχουν μια εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των ε, τελωνιακών ε, αρχών. Κατά την άποψή μου θα πρέπει οι δαπάνες εδώ να μεθούν από 20% στο 10%. Ε, το 20% ήταν έμεσες ε, εισπράξεις για τις χώρες μέλη, όπου πραγματικά γίνεται το σημαντικό εμπόριο. Με 10% καλύπτονται οι δαπάνες για το Ρότερταμ, για το Αμβούργο ή για την ε, Γένοβα ή για την Αμβέρσα. Με 20% οι χώρες της μέλη έχουν ένα κίνητρο για να διεξάγουν τους ελέγχους. Άρα το 10% είναι αντικειμενικά ερθό, αλλά ίσως δεν είναι ιδιαίτερα έξυπνο. Ε, έξυπνος ο ορισμός αυτού του ποσοστού γιατί δεν παρέχει επαρκή κίνητρα. Αναμένουμε την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου όσον αφορά το ΕΦΣΥ. Εδώ έχουμε τις ε, ε, εισφορές των νέων χωρών, έχουμε ανάλυση κόστους εφέλειας κλπ. Ε, και είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε σοβαρά το, τις ε, συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Αλλά εδώ δεν υπάρχουν σταθερά μερίδια των χωρών ε, μελών, ε, γιατί το ζούμενο είναι η καταλληλότητα αλλά και η υψηλή ποιότητα των χωρών. Και είναι πολλές χώρες οι οποίες δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν, ενώ άλλες είχαν έντονο ενδιαφέρον να ε, συμμετάσχουν εδώ ε, στο πρόγραμμα ε, Juncker. Θα, θα προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε τις τάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου ε, τους πρώτους μήνες του προσεχούς έτους. Τώρα, ε, πρόεδρος, όσον αφορά για την μία αξιοποίηση των ε, πληροφοριών, απαντήσατε ότι ε, πρόκειται για στοιχεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο εκ των εξτέρων. Θεωρώ ότι δεν μας καλύπτει η απάντηση. Η έκθεση αυτή πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μας. Ο, οι συνάδελφοι, ο κύριος Σάβαμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, καλά τα καταφέρατε. Ε, χαιρόμαστε πολύ που είσαστε εδώ, κύριε Επίτροπε και εσείς. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε ορισμένα σημεία ως προς την εκτενή αυτή συζήτηση. Δεν νομίζω ότι κανένα σας ευχαρίστησε για την έγκαιρη κίνηση της ε, περίοδου διακοπών Ε, όμως ε, δεν πρόκειται για διακοπές ως προς την δημοσιονομική διαδικασία. Εν πάση περιπτώσει έχουμε ξεκινήσει με μια διαδικασία πανηγυρικών εκδηλώσεων. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα υπόλοιπα προς εκαθάριση, για τα ραλ. Να και πάλι, στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε. Το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι πρέπει να γίνει πλέον. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα χάσματα πληρωμών που συσσωρεύονται στο τέλος κάθε πολιετούς. Τώρα, ως προς τις κεφαλίδες, ε, στην ε, κεφαλίδα 1 υπάρχει ένα σαφές μήνυμα προς την Επιτροπή σε σχέση με τα μη επιλέξιμα, τις ε, μη επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνουν οι δικαιούχοι. Άρα κάτι είναι λάθος στην όλη διαδικασία ελέγχου. Με τα ποσά που βλέπουμε, τα οποία είναι σχετικά υψηλά ως προς το, τις μη επιλέξιμες δαπάνες ε, που υπησέρχονται. Τα δύο μεγαλύτερα κεφάλαια είναι η ΚΑΠ και η συνοχή. Για την ΚΑΠ θα ήθελα να πω ότι όταν δω το συνολικό επίπεδο σφάλματος 2,4, ξέρουμε ακριβώς ε, τι αφορά Θέλουμε όμως λεπτομέρειες γιατί στο δεύτερο πυλώνα και στην αγροτική ανάπτυξη παραμένει πολύ υψηλό το ποσοστό σφάλματος. Ποια είναι η πραγματική εικόνα. Δεν είναι σαφής, δεν είναι απόλυτα σαφής για τα μέλη της ε, Επιτροπής μας και θα πρέπει να δούμε λεπτομερώς αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Ως προς τη συνοχή τώρα, Έχω ένα ερώτημα και εδώ, γιατί δεν κατανοώ πώς φτάνουμε στο συμπέρασμα ή μάλλον ε, ας το επαληθεύσουμε, ας το ελέγξουμε καλύτερα. Λέτε ότι το 3,0 το ποσοστό σφάλματος οφείλεται στα χαμηλά ποσά, ποσοστά αποδεκτών δαπανών, τα 8 δις δηλαδή, γιατί δεν καταλαβαίνω πώς ε, επιδρά τόσο πολύ στο ποσοστό σφάλματος. Επίσης, Προς το τέλος του δημοσιονομικού πλαισίου θα αυξηθεί το ποσοστό για το 2018. Πώς επιδρά στο σφάλμα καθεαυτό, στο ποσοστό σφάλματος. Και κάτι άλλο για το EDF. Εάν κατανοώ σωστά, επειδή Επιτροπή οποίοι έχει ευελιξία σε σχέση με την ε, προκριματικότητα και επειδή δεν γίνεται σωστή χρήση των εθνικών κονδυλίων, δεν μπορεί να αναγνωριστεί σωστά το σφάλμα. Δηλαδή από το 3,3 περνάμε στο 2,5 παρά το γεγονός ότι υπησέρχονται έλεγχοι. Και έχουμε να κάνουμε βεβαίως και με, τρίτα, και με τρίτους σε επικίνδυνους τομείς όπως είπε και ο Επίτροπος Έτιγκερ. Τι θα γίνει όμως με το ποσοστό σφάλματος ως προς το διορθωτικό προϋπολογισμό. Τα ίδια λέω χρόνο με το χρόνο, αλλά χρειάζεται διαφάνεια ως προς αυτές τις δαπάνες. Διαφορετικά, ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού δεν θα είμαστε σε θέση να πούμε πού και πώς κατασπαταλούνται τα ε, χρήματα. Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ. Κύριε Λένε, κύριε Επίτροπε, μετά από τις διάφορες παρεμβάσεις, ας έρθουμε σε κάποια αρνητικά της ε, τρέχουσας κατάστασης. Θα προσπαθήσω να αξιολογήσω τα τέσσερα της συνεργασίας μας με τον Επίτροπο Έτιγκερ. εδώ, στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Λοιπόν, σημειώθηκε πρόοδο όλα αυτά τα χρόνια. Το ποστό σφάλματος μειώθηκε και, και ως ποσοστό, αλλά νομίζω και σε απόλυτους όρους. Είναι σημαντικά και τα απόλυτα μεγέθη. Δεύτερον, συμφωνήσαμε σε μεγάλο βαθμό ότι κοινός μας στόχος είναι να μεγιστοποιήσουμε την λεγόμενη προστιθεμένη αξία, το υπογράμμισε αυτό και ο πρόεδρος Λένα. Εμείς θα περιμέναμε, οφείλω να ομολογήσω, μια καλύτερη κατανομή των κονδυλίων και υψηλότερη επίδοση, υψηλότερη απόδοση στην αξιοποίηση των κονδυλίων. γιατί αυτό θα ήταν καλό για την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μη αξιοποίηση, η κακή αξιοποίηση, για μένα σημαίνει ότι καλύτερο θα ήταν να μην είχαμε στείλει καθόλου εκεί τα κονδύλια. Γιατί αλλιώ γίνονται λάθη, έχουμε περιστατικά απάτης κλπ. το λέω αυτό και για το 18 αλλά και το, για το δεύτερο εξάμεινο του 17. Και το λέω διότι εκκρεμούν όλο και μεγαλύτερα ποσά σε πιστώσεις πληρωμών. Ανοίγει το χάσμα δηλαδή μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι εν τέλει καλό. Ας πούμε για την Πολωνία για παράδειγμα. παρά το γεγονό ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε το 1,5 2% τη ετήσιας ανάπτυξή μα στην Πολωνία. Και ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουν όντω για ανάπτυξη. Χρειάζεται επίσης περισσότερη διαφάνεια και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής κανόνων, περισσότερων κανόνων. Αυτό όμως μπορεί να είναι και αντιφατικό. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι το βέλτιστο επίπεδο κανόνων και κανονισμών. Να συγκρίνουμε πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, να δούμε ποια είναι η χρυσή τομή. Κάτι άλλο που ήταν καλό αυτά τα τέσσερα χρόνια ήταν αυτό που είπε και ο πρόεδρο Λένε, ότι δηλαδή έχουμε αρκετή ευελιξία, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερη. Διαπιστώσαμε επίσης ότι η κατανομή των κονδυλίων πρέπει να γίνεται με πιο, πάνω σε πιο ρεαλιστική βάση. Να απέχει λιγότερο η θεωρία από την πράξη, από αυτό το οποίο προκρίνεται τελικώς. Εν γέννη πιστεύω ότι τα τέσσερα τελευταία χρόνια ήταν καλά, έγινε νομίζω σωστή δουλειά. Αποδείξαμε ότι δεν είμαστε υπερόπτες. Δουλεύουμε, έχουμε πολλά μπροστά μας Οπότε κλείνω ευχαριστώντας το Ελληνικό Συνεδρίο και τον Επίτροπο. Η δουλειά στην Επιτροπή μας θα συνεχιστεί. Ε, λοιπόν, πρέπει να φύγω λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ε, μίλησαν με τόσο φιλικά λόγια. Κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι αυτό το οποίο εμεί ανακαλύψαμε θα μπορούσαν να είχαν ανακαλύψει και άλλοι. Τότε διαρωτώ με, γιατί δεν το έπραξαν. Και μια άλλη ερώτηση. Το μέλος του Αυτακού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Χέριτς, έδωσε χτες μια ε, ε, ανακοίνωση τύπου. Εμείς πήραμε την ε, έκθεση χτες στα χέρια μας. Είναι αποδεκτό κάποια μέλη να απευθύνονται στην δημοσιότητα με τον τρόπο αυτό. Τώρα, για τον Επίτροπο κύριο Έτεγκερ. Θεωρώ ότι είναι πολύ θαραλέα η δήλωσή του ότι Επιτροπή ε, λαμβάνει υπόψη της ε, με, ε, ήδη στη βάση μιας πλατιάς συμφωνίας την έκθεση. Ή το ποστό σφαλμάτων δεν οφείλεται σε απάτη. Ή θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την συμβατότητα των εργαζομένων. Δεν ξέρω, γιατί αναφέρεται στην έκθεση του ΕΝΤΕΕΦ ότι ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, με πρόθεση ε, η Επιτροπή δεν, δεν διεξήγαγε σωστά ε, ορισμένους ε, ελέγχους που αφορούσαν όμως ε, αρκετά μεγάλα ποσά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πραγματικά δίνουν λαβή για σοβαρές σκέψεις. Επίσης, όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, εγώ ε, θεωρώ ότι δεν πρόκειται για το σχέδιο Μάρσαλ εδώ και πραγματικά ε, είναι δύσκολο να διεξαχθεί εδώ κάποιος έλεγχος. Θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα όσον αφορά αυτά αυτή τη βοήθεια. Τώρα, οι συστάσεις ε, που έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο το 2014 προς την Επιτροπή 58% ε, υλοποιήθηκαν, 6% καθόλου. Γίνεται ετήσια ένας έλεγχος εν σχέση με το πώς υλοποιούνται οι συστάσεις. Γιατί εγώ θα θεωρούσα ότι θα πρέπει να γίνεται αυτό εν πάση περιπτώσει, γιατί οι συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου έχουν μεγάλη βαρύτητα, αλλά θα έπρεπε κατεπηγόντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβαίνει στην ε, υλοποίησή τους. Όχι να λέει ότι απλώς τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη της συμφωνώντας ως προς τα περισσότερα σημεία. Τώρα, όσον αφορά τις εσμεύσεις των κονδυλίων, εγώ ε, ε, είχα κάνει μια πρόταση στην Επιτροπή να, υπάρξει, να απελευθερώσει κάποια κονδύλια για, στο πλαίσιο κάποιων ε, επίκαιρων ε, αναγκαιοτήτων. Ε, και μου είπαν ότι δεν γίνεται, έχουν ήδη δεσμευτεί τα χρήματα αυτά. Εγώ θεωρώ θα πρέπει να έχουν κάποια ευελιξία, όχι να δεσμεύονται αρχικά τα χρήματα και μόνο να γίνονται οι επιστροφές τέλος του έτους και τελικά τα χρήματα αυτά να καταλήγουν, να γίνονται άχρηστα, να θα τα είχαμε χρειαστεί για πολύ πιο σημαντικά ζητήματα. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σε αυτό το όψιμο στάδιο θα είμαι σύντομος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να ανησυχούμε ιδιαίτερα με τα στοιχεία αυτής της έκθεσης και νομίζω ότι υπάρχουν τρεις λόγοι γι' αυτό. Το θέμα της απορρόφησης, κανονικότητας και αποτελέσματος. Αν ε, μιλήσουμε για την απορρόφηση, όλοι αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι οι υποχρεώσεις έχουν αυξηθεί δραστικά. Έχουν φτάσει σε ένα ποσοστό ρεκόρ και ο συνολικός ε, ρυθμός απορρόφησης του 16% είναι πολύ υψηλότερος από ότι στο αντίστοιχο δημοσιονομικό πλαίσιο που ήταν 22%. Ε, Άρα το συνέδριο μας το επεξήγησε γιατί έκλεισε αργότερα το προηγούμενο πολιετές ε, είχαμε νομοθετήματα πολύ πιο αργά και αλλαγές ως προς την απαλλαγή εν συν 2, νη συν 2 και νη συν 3 και φυσικά για τα κενά που υπήρξαν στα, στο προηγούμενο πολιετές. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε αγκιστρωθεί σε αυτή την ε, εικόνα και είναι ακόμα και πιο δύσκολα τα πράγματα ως προς την κανονικότητα και τα δημοσιονομικά μέσα. Ακούσαμε από τον Επίτροπο ότι μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά, τα οποία μπορεί να είναι και βάλτος. Μπορεί να βαλτώσουμε τελικά. Είναι δύσκολη πλοήγηση τα δημοσιονομικά μέσα. Ε, συνεισέφεραν στο ποσοστό σφάλματος και υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Ποιος ευεργετείται από τα δημοσιονομικά μέσα. Ε, δεν υπάρχουν ποσοστώσεις για τις μεμονωμένες χώρες. Πού θα πάνε τα χρήματα λοιπόν αυτά. Ως προς την συνοχή οικονομική και κοινωνική καθώς και εδαφική συνοχή βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών και περιφερειών και νομίζω ότι αυτό θα είναι αποφασιστικό για την τύχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή κατά πόσο οι ανισότητες θα αντιστραφούν και θα αρχίσει να λειτουργήσει η συνοχή ή όχι. Και ό,τι, απομείνει αυτή, ό,τι απομένει από αυτή την έκθεση είναι η οχι και οτι αυτη οτι απομενει απο ότι δεν θα υπάρξει σύγκληση. Είχαμε οκτώ δις ε, στη συνοχή. Αυτές ήταν οι δαπάνες. Και ε, υπήρξε ένα ποσοστό μη ελέγχου σε σχέση με αυτά τα 8 δις. Αυτό φυσικά σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα το 18 και 19. Άρα θα υπάρξει μία συσσόρευση σε αυτές τις χρονιές. Τώρα, ως προς τα αποτελέσματα, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σημαίνουν ε, επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Άρα θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις για να δούμε κατά πόσο επιτυγχάνονται αυτά τα, αυτοί οι στόχοι. Εδώ θα πρέπει να καλύψουμε πολύ έδαφος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προσέξουμε αυτή την έκθεση, να δούμε ποια είναι τα ευρήματα και φυσικά τις συστάσεις που προέβαλε το ελεγκτικό. Αλλά θα ήθελα να καλέσω όλους να μην χάσουμε το δάσος εξαιτίας ε, των δέντρων. Δηλαδή, η συνολική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Θα είμαι σύντομο. τρει παρατηρήσει. Πρώτον, Προ την Κομισιόν. Η οποία πρέπει να επενεθεί. Σημείωσε σημαντική πρόοδο. Φαίνεται άλλωστε αυτό και στην έκθεση που συζητούμε. Όλα αυτά χάρη στην Κομισιόν, χάρη στο προσωπικό, τα στελέχη, το άλλο, το προς εκταμείευση υπόλοιπο, τα ραλ. Βεβαίως, αναγκαστικά έτσι διαχειρίζεται κανείς επενδύσεις, όμως το ύψος των ραλ πρέπει να την χάνει επαρκούς διαχείρισης. Εμπροκειμένου να επενθυμίσω στην Κομισιόν ότι στον περασμένο προπολογισμό είχαμε θέσει πολύ συγκεκριμένο στόχο για την διατήρηση και μάλιστα την μείωση του ύψους των ραλ και η Κομισιόν σημείωσε εκεί σημαντική πρόοδο. Διαχειρίστηκε και τα μείωσε. Για μένα, όπως και για άλλους συναδέλφους, είναι ενισχυτικό ότι η τάση αυτή αναστρέφεται όχι μόνο επιβραδύνθηκε, αλλά και αναστρέφεται. Και εδώ κύριε Πρόεδρε έχουμε πράγματα να συζητήσουμε. Κύριο Τρίτο, συγγνώμη επαναλαμβάνομαι, γινόμαστε πληκτικοί για τον Πρόεδρο του Ελληνικού Συνεδρίου, αλλά η έκθεση είναι ευκαιρία να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στο ευρύ κοινό να καταλάβει ο κόσμο ότι υπάρχει αποτελεσματικό έλεγχο του προπολισμού. Και αυτό μπορεί μόνο να εξασφαλιστεί με λογοδοσία και διαφάνεια. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποια θέματα είναι λεπτά. Το έχουμε συζητήσει αυτό και στο παρελθόν. Όμω, επιτρέψτε μου να πω και πάλι ότι όσο περισσότερα στοιχεία, όσο καλύτερα στοιχεία, όσο πιο αξιόπιστα στοιχεία δίνουμε με παραδείγματα, με λεπτομέρειες, με συγκρίσεις στην έκθεση, τόσο καλύτερα. Έτσι εξασφαλίζουμε την διαφάνεια, άρα όπως είπα εμπιστοσύνη στο κοινό, αλλά και για μας ξέρετε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Είναι ένα μέσο να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτεραιότητες στον τομέα των επενδύσεων. Ο Σέντρος Κούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαζάρ, κύριε Επίτροπε, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ ότι είναι ένα μέσο το οποίο μπορούμε να το πουλήσουμε θετικά προς τους Ευρωπαίους πολίτες, ότι, έχουμε ένα... ότι το ποσοστό σφαλμάτων υποχωρεί. Και νομίζω ότι παρά τις αρνητικές παρατηρήσεις, αυτό είναι το βασικό θετικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να... στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα. Τώρα, εγώ είμαι συγητής για τα άλλα θεσμικά όργανα και στον τομέα της διοίκησης. Έστω και αν σε χαμηλό επίπεδο, εδώ βρισκόμαστε σε ένα διπλασιασμό του ποσοστού σφάλματος. Ε, θα ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα. Και ένα, μια διευκρινιστική ερώτηση, σελίδα 7, είναι οι δεσμεύσει ε, ε, κονδυλίων που θα πρέπει να γίνουν, που εκκρεμούν ε, εδώ το καταλαβαίνω καλά, πρόκειται για προγράμματα τα οποία βρίσκονται υπό εξέλιξη, κονδύλια για τα οποία δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει τα προγράμματα. Τι εννοείται με αυτό. Ε, θα ήθελα να καταλάβω τι εκκρεμεί ακόμα. Ε, είναι γενικά, εκκρεμούν γενικά τα προγράμματα ή εκκρεμεί η πληρωμή. Ο κύριος ε, Τσέλερ, ευχαριστώ πολύ και εγώ από την πλευρά μου, κύριε Ελένη, κύριε Λαζάρου, ξέτοιμα μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο κύριο Έτιγκερ για τις πληροφορίες όσον αφορά την ε, ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι μια βάση της εργασίας μας, όπως και, τα, όπως και οι εκθέσεις των ε, Γενικών Διευθύνσεων. Ε, πολλοί συνάδελφοι είπαν ότι τις άμεσες πληρωμές έχουμε όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος είναι, έχουμε μια ελαφρά βελτίωση εδώ. Αλλά πιστεύω εδώ βρισκόμαστε σε ένα τομέα όπου δεν θα μπορέσουμε να επιφέρουμε περαιτέρω βελτιώσεις. Γιατί ε, ε, συνήθως έχουν γίνει διορθώσεις και λοιπά. Άρα συνήθως είναι 2% το ποστό των σφαλμάτων. Ε, επίσης πρόκειται για σφάλματα επίσης στην διαδικασία ε, ε, ε, ανάθεσης των δημοσίων έργων. Εκεί γίνονται τα περισσότερα σφάλματα. Η σχετική οδηγία εκδόθηκε το 2014 από την ε, Κομισιόν και στις περισσότερες χώρες δεν έχει εφαρμοστεί. Σε ορισμένες με καθυστερήσει, σε άλλες καθόλου ε, και υπάρχουν πολλές παραβιάσεις στη διαδικασία ανάθεσης ίσως θα έπρεπε να το δούμε αυτό για να υπάρξει μια περαιτέρω μείωση στο, του ποσοστού σφαλμάτος. Αυτό θα έπρεπε να μας βάλει σε θέση να δούμε και τους τομείς εκείνους όπου πραγματικά ε, διερωτώμαθα κατά πόσο έχει επιτευθεί η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Την περασμένη εβδομάδα μιλήσαμε για τα τρένα υψηλής ταχύτητος. Οι χώρε μέλη έφτιαξαν το σχετικό σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά όλα στο εσωτερικό του σιδηροδρομικό δίκτυο και εκεί που θα έπρεπε να παραχθεί η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία, δηλαδή διασυνοριακά, Εκεί δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Συνήθως ε, λίγοι σταματάει το δίκτυο 20 χιλιόμετρα πριν από τα σύνορα. Ίσως θα έπρεπε εδώ να κάνουμε κάποια κριτική και να προσέξουμε τα κονδύλια τα οποία έχουν διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι να πετυχάνουν τη λεγόμενη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ε, και μη ικανοποιητική, και συμφωνώ με τον κύριο Σβίτ, είναι μη ικανοποιητικό στον τομέα η Ευρώπη στον κόσμο και η αναπτυξιακή συνεργασία. Ε, τα όσα αναφέρει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου με κάνουν να συμπεράνω ότι το ελεγκτικό συνέδριο παρετείται από αυτή την προσπάθεια διότι λέει δεν είναι δυνατός ο έλεγχος εδώ και μάλιστα σε ένα τομέα που πραγματικά ε, χρειαζόμαστε κατεπηγόντως ε, έναν ε, έλεγχο και μια εκτίμηση η οποία να προσανατολίζεται ακριβώς τα αποτελέσματα. Πόσα χρήματα φεύγουν το output όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο περίπου 12 δις αλλά δεν βλέπουμε ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί. Βλέπουμε πόσα χρήματα έχουν φύγει, αλλά τι έχει ε, επιτευχθεί στην πράξη δεν το ξέρουμε. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω εδώ να δοθεί μια προτεραιότητα τόσο όσον αφορά την εργασία του ελεγκτικού συνεδρίου όσο και των αρμοδίων επιτρόπων. Δεν είναι απολύτως αποδεκτό αυτό το οποίο πρόεδρό μας Ε, δηλαδή ότι οι αιτήσεις εκθέσεις των ευρωπαϊκών αντιπροσωπιών ε, δεν γίνονται, δεν ε, συζητούνται και κλεισμένων των θυρών, αλλά δημοσία. Σε ασμένες από αυτές, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων με τα κονδύλια μας, ε, στέκονται σε πολύ σαθρά πόδια. Τα περισσότερα ε, χρήματα πάνε σε συνεργασία με οργανισμούς των Ηνωμένων Αθηνών, ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας κλπ. Δηλαδή, ε, τα αποτελέσματα της, αναπτυξιακής, της χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας δεν είναι ορατά στις ίδιες τις υποανάπτυξη χώρες, αλλά τα μοιράζονται οι διάφοροι οργανισμοί μεταξύ τους. Ε, και το να είναι ορατή η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο μέσω των αντιπροσωπιών που μεταβαίνουν σε μια χώρα και βάζουν τη σημαία τους, ε, θεωρώ ότι είναι ανεπαρκές. Ο κύριος Έτιγκερ είχε πάει την περασμένη εβδομάδα στη, στα Έθνη στη Νέα Υόρκη ε, τους πρόεδρους των επιτροπών ε, εκεί ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια πράγματα σχετικά και Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπούλα. Uh, uh, uh, Ευχαριστώ. Το πρώτο θέμα που θα ήθελα να τονίσω είναι η, η ουδετερότητα και αμεροληψία του ελεγκτικού συνεδρίου. Από ό,τι φαίνεται, η, τα μέλη είναι κατά 40% πρώην πολιτικοί καθώς και ανώτεροι αξιωματούχοι των ε, θεσμικών οργάνων, 45% του προσωπικού. Πρόκειται για σύγκρουση συμφέροντος. Θα πρέπει να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη και να δείτε το νομικό ορισμό της, ε, του θέματος. Με ανησυχούν τα στοιχεία σε σχέση με μεμονωμένες ε, περιπτώσεις γιατί πέρσι είχαμε τα ακριβή ε, project για κακή δαπάνη. Ε, φέτος τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα ασαφή. Υπάρχει αδιαφάνεια και αυτό νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Ένα άλλο σημείο που με κάνει να αμφισβητήσω την αρμοδιότητά σας είναι ο δικός σας προϋπολογισμός. Μιλάμε για 45.000 ευρώ που δαπανήθηκαν για την 400η επέτειο του ελεγκτικού. Και ε, πρόσφατα δαπανήθηκαν γύρω στις 100 ε, με 150 για επιμέρους ε, πανηγυρισμούς και εκδηλώσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για 166 δις και ζημία της τάξης των 36 ε, δις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης είχαμε ένα τέτοιο θέμα στο Northampton και το Δημοτικό Συμβούλιο στην ουσία χρεοκόπησε και ε, στάλησαν κρατική λειτουργή για τη διαχείριση. Στη σελίδα 10 μιλάτε για την νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών πίσω από τους λογαριασμούς. Όμως, εάν ένας επιχειρηματίας στον ιδιωτικό τομέα λάμβανε αυτά τα στοιχεία, θα ήταν προβληματικά. Μιλάτε επίσης για 2,4% δηλαδή 4 δις ευρώ του χρήματος του φορολογούμενου που δεν έχει δαπανηθεί σωστά. Υπάρχουν πολλοί όροι, πολλά caveat που ε, αναφέρονται και επίσης μας απασχολεί και το μέγεθος του δείγματος σε ορισμένους ελέγχους. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Στην κεφαλίδα 3 σε σχέση με την ασφάλεια και την ε, ηθαγένεια δεν υπάρχει ποσοστό σφάλματος. Στη σελίδα 333 αναφέρεται ότι οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου, άρα δεν έχουν επέλθει σφάλματα. Αυτό είναι γελίο. Επίσης, αυτή η έκθεση μιλά για παράβαση και κατασπατάληση χρήματος εκεί που υπάρχουν σφάλματα. Όμως έχουν υπάρξει πολλές δαπάνες οι οποίες δεν είναι καθόλου ε, σκόπιμες. Γι' αυτό πρόκειται για κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Ευτυχώς που το Brexit για μας σημαίνει ότι δεν θα συνδράμουμε σε αυτή τη διαδικασία στο μέλλον ή τουλάχιστον αν συνδράμουμε θα είναι απειροελάχιστα. Ε, διαβάσατε αυτό το οποίο σας είχαν ε, γράψει το ένα τρίτο ήταν σωστό. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ στο περαιτέρω. Ναι. Κύριος Τσαρνέσκη έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Οι προλαλήσαντες είπαν σοφά πράγματα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω το Ελληνικό Συνέδριο για την έκθεση, η οποία φέρος υποβάλλεται νωρίτερα και αυτό βεβαίως είναι θετικό. Θέλω επίση να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε. Τα φετινά αποτελέσματα όμως επιβεβαιώνουν τα ευρήματα περασμένων ετών. όσον αφορά τον τρόπο δαπάνης των κονδυλίων, ε, όσον αφορά τις επιπτώσεις από τα σφάλματα, καθώς και όσον αφορά τις δαπάνες που εκταμιεύονται με βάση δικαιώματα. Σε αυτά τα προγράμματα, στα τελευταία αυτά προγράμματα, το το σφάλματος είναι υψηλότερο. Και φαίνεται επίσης ότι το σφάλμα είναι υψηλότερο εκεί όπου τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι πιο πολύπλοκα. Άρα εκεί πρέπει να εστιαστούμε, να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε την ποιότητα των εκθέσεων σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων. Εκεί δεν μας δίνουν αρκετά στοιχεία. Πολλά είναι απλώς εκτιμήσεις για μελλοντικές δαπάνες. Γενικά πάντως τα πήγατε καλά νομίζω και ευχαριστώ πολύ. Α, με συγχωρείτε. Ε, ο συνάδελφος, ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδίνετε την ευκαιρία να προσθέσω κάτι που ξέχασα γιατί ήμουν υπερβολικά επικεντρωμένο στα προηγούμενα που είπα και παρασύρθηκα. Λοιπόν, Δεν μπορώ να πω ότι είναι και η καλύτερη μέρα, ότι είναι και γιορτή σήμερα για τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο. Αλλά την ημέρα έκδοση λοιπόν της έκθεσης πρέπει να ευχαριστούμε τον κύριο Λαζάρου, τον αναντικατάστατο ε, συνοδοιπόρο του κυρίου ε, Λένε, χωρίς τον οποίο δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λαζάρου. Κύριο Λαζάρου. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ερωτήσεις σας και να ευχαριστήσω και τον κύριο Σαββαμά για τα καλά του λόγια. Η δύση έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. Οπότε, μέσω εμού, μέσω του Προέδρου και εμού, πιστεύω ότι τα καλά λόγια πρέπει να μεταφερθούν και ταξίζουν τα στελέχη μας και το προσωπικό του ελεγκτικού συνεδρίου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω εν συνεχεία να απαντήσω όσο πιο καλά μπορώ στις ερωτήσεις σας. Και εν συνεχεία ο πρόεδρος εφώς θα συμπληρώσει και θα ολοκληρώσει. Κύριε Σαβαμά, αμφισβητήσατε τη γενική εικόνα στον αφορά τη γεωργία. Δεν κατάλαβα, ομολογώ, την ουσία της ερώτησης, όμως εντάχει να σας ενημερώσω για τα εξή. Στην ε, Γεωργία, γενικώ το ποσοστό σφάλματος ήταν 2,4. Αυτό αφορά τις άμεσες ενισχύσεις από το Γεωργικό Ταμείο, καθώς και τα μέτρα για την αγορά. Στην ετήσια έκθεση διευκρινίζουμε επίση ότι στις αμέσες ενισχύσεις το ποσοστό σφάλματος είναι κάτω από το κατόφλι σημαντικότητας. Συνολικά το ποσοστό είναι 2,4% όπως είπα. Δεν έχουμε για τη γεωρική ανάπτυξη αντίστοιχο ποσοστό, για τα μέτρα γεωρικής ανάπτυξης, ε, όμως ε, καταλαβαίνετε ότι θα είναι υψηλότερο του 2,4% δεδομένου ότι έχει, έχουν σταθμιστεί δύο πυλώνες. Άρα, βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, όσον αφορά τη γεωργία και όσον αφορά το Ταμείο Συνοχής. Φέτος, τα αποδεκτά κονδύλια ήταν μόνο 8 δισεκατομμύρια. Αυτό ελέγξαμε. 8% του επιλέξιμου για έλεγχο δαπανών. Το 2016 τα αντίστοιχα κονδύλια ήταν σχεδόν 36 δισεκατομμύρια. 28% του συνόλου των δαπανών. Το 2016 στη συνοχή το ποσοστό ήταν 4,8% το ποσοστό σφάλματος και φέτος πιθανότερα θα κινηθούμε γύρω στο 3%. όταν λέω το πιο πιθανό, ε, αυτό δεν συναρτάται με το ποσό των αποδεκτών δαπανών. Υπάρχει σχέση βεβαίω μεταξύ των δύο, όμω η συμβολή τη συνοχή το 2017 στο συνολικό σφάλμα είναι, για του λόγου που εξήγησα, χαμηλότερη σε σχέση με το 2016. Γιατί τότε ήταν η συνοχή 28%, ενώ ε, φέτο έχουμε μόνο 8 δισεκατομμύρια και 8% αντίστοιχα συμπτωματικά. Αυτό εξηγεί και την μείωση του συνολικού ποσοστού σφάλματος από το 2016 στο 2017 από 3,1 στο 2,4. Βεβαίω, εν τω μεταξύ έγιναν και άλλες βελτιώσεις, όμως μέρος αυτής της διαφοράς εξηγείται ακριβώς από τη συμμετοχή, του σχετικό βάρος δηλαδή των δαπανών του Ταμείου Συνοχής. Τώρα για το Ταμείο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Και Πάλι εκεί με ρωτήσατε ποιο είναι το ποσοστό συμμετοχή. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σα. Να πω όμω εν γέννη ότι για το EDF έχουμε ξεχωριστή ετήσια έκθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες ε, θα διαβάσετε στην ετήσια έκθεσή μας. Και να προσθέσω ότι το ανώτερο ποστό σφάλματος 7,8% και το χαμηλότερο 1,2%. Μέσος όρος 4,5%. Όσον αφορά όμως, όπως είπα, τη συμβολή του τομέα στο συνολικό σφάλμα, όχι, το μειώνει γιατί επειδή πηγαίνουν στον εθνικό προπολογισμό δεν υπάρχει σφάλμα εκεί επειδή όμω συμμετέχουν οι δαπάνε στο σύνολο των δαπανών, το αποτέλεσμα είναι το συνολικό σφάλμα να μειώνεται. Κύριε Σμιτ, ρωτήσατε εάν οι συστάσεις των περισμένων ετών λαμβάνονται υπόψη και υλοποιούνται. Ναι, κάθε χρόνο διαβάζουμε τις ε, συστάσεις των τελευταίων τριών ετών, ας πούμε στο κεφάλαιο 3 επιδόσεις, ανατρέξαμε στις συστάσεις του 14. Οι περισσότερες από αυτές έχουν υλοποιηθεί, ε, αλλά και για τα επιμέρους κεφάλαια. Έχουμε έναν πίνακα στο παράρτημα, όπου αποτυπώνονται οι συστάσεις τρία χρόνια πριν και περιγράφουμε που ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τρία χρόνια μετά το έτος δηλαδή της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης. Κύριε Κόν, θέσετε μια ερώτηση αν υπάρχει μια τάση στο κεφάλαιο 5 του η διοίκηση και γιατί μειώσαμε τον αριθμό των συλλαγών. Και επίσης ε, ζητήσετε μια εξήγηση όσον αφορά την σελίδα 17 όσον αφορά τις εκκρεμείς πιστώσεις υποχρεώσεων. Στον τίτλο, κοιτάξτε, 5 δεν υπάρχει τάση. Ή, να το πω αλλιώς, η τάση είναι ότι ούτως ή άλλως το ποσοστό είναι κάτω από το 2%. Είμαστε κατά κόρον κάτω από το 2%. Είμαστε συνεχώς κάτω από το 2% και όταν το ποσοστό είναι ε, τόσο χαμηλό, τότε δικαιούμεθα να μειώσουμε το δείγμα. Γιατί θεωρούμε ότι σύμφωνα με τα πρότυπα έχουμε αρκετέ πληροφορίε για να καταλήξουμε σε γνώμη. Γνώμη ελεγκτή. Για την ε, 17, ο έλεγχος εν συντομία, περιγράφουμε τις εκκρεμείς πιστώσεις υποχρεώσεων ανά κράτος μέλος όσον αφορά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Και λέμε που βρισκόμαστε μέχρι στιγμή. Αυτό είναι που συζήτησαμε και προηγουμένω. Τώρα, δεξιά στη σελίδα αυτή διαβάζετε τα ποσοστά αυτών των εκκρεμουσών πιστώσεων δεσμεύσεων σε σχέση με τις κυβερνητικές δαπάνες. Ανακρατός μέλος. Είπατε για την ε, ουδετερότητα και την αμεροληψία του ελεκτικού συνεδρίου, διότι δουλεύουν σε εμά πολιτικοί, δημοσιοί πάλι κλπ. Και αμφισβητήσατε την ε, με σχόλια γνώμη και είπε ότι μια ιδιωτική εταιρεία αντίστοιχα δεν θα ήταν ε, ικανοποιημένη με την κανονικότητα και νομιμότητα στο σημείο που έχουμε φτάσει. Εγώ θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Πούλοκ και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού περί της ουδετερότητας και αμεροληψίας αλλά και περί του επαγγελματισμού των μελών του Ελεκτικού Συνεδρίου. Νομίζω ότι η ουδετερότητά μας είναι αναμφισβήτητη, δεσμευόμεθα από διεθνή πρότυπα, από κώδικα δεντολογίας και διενεργούμε τους ελέγχους μας σύμφωνα με τα πρότυπά μας και τις αρχές μας. Μας υποστηρίζουν περίπου 900 επαγγελματίες, 900 στελέχη, είναι όλοι τους επαγγελματίες και συμμορφώνονται με τη βίβλο μας, δηλαδή τα πρότυπα, κάνουμε τη δουλειά μας επαγγελματικά, ακριβώς όπως θα την έκανε ένας οποιοδήποτε ιδιώτης εξωτερικός ελεγκτής. Τώρα, για τη γνώμη με σχόλια. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θετικό βήμα, γιατί επί πολλά χρόνια είχαμε αρνητική γνώμη για κανονικότητα και νομιμότητα. Από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχουν πολλές ελεγκτικές αρχές στα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διενεργούν ελέγχους συμμόρφωσης και που δίνουν όλα αυτά τα στοιχεία συμπεριλαμβανομένου και του ποσοστού σφάλματος. είμαστε σε θέση να εκτιμούμε τη συμμόρφωση. Αυτό γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκπρόσωπος του Εθνικού Γραφείου Ελέγχου ήταν στο Κοινοβούλιο πριν από καιρό και είπε όταν απαντούν σε σχετική ερώτηση όσον αφορά το ποσοστό σφάλματό του. Και πρέπει να σα πω ότι στην Αμερική, στι ΗΠΑ, το ποσοστό σφάλματό του είναι πολύ ψηλότερο από αυτό το οποίο έχουμε καταγράψει εμεί στην σημερινή μα έκθεση. Εν πάση περιπτώσει, δεν θεωρούμε ότι είναι κακό μια γνώμη με σχόλια. Ίσα ίσα περί του αντιθέτου πρόκειται. Ευχαριστώ. Στι Ηνωμένε Πολιτείε το ποσοστό σφάλματο είναι 10%. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει τώρα να, να μιλήσω με κάπως γενικότερους όρους. Ο κύριος Κούνη είπε ότι θα πρέπει να του εξηγήσουμε τι είναι αυτό το ποστό σφάλματος. Θα ήθελα να πω το εξή. Δεν είμαστε σε θέση ε, κάθε διαδικασία που έχει λάβει η χώρα στην, ε, να την ελέγξουμε. Έχει, ε, έχουμε έξι εργαζόμενους στο τομέα του ελέγχου και ε, μπορούμε να τα κάνουμε, κάνουμε τους ελέγχους αυτούς άρα μόνο δειγματοληπτικά. Σαν μια δημοσκόπηση ε, ρωτούνται οι άνθρωποι για την άποψή τους και στη συνέχεια αναλυτές της κοινή γνώμης ορίζουν κάποια, καταλήγουν σε κάποια ποσοστά. Αλλά μπορεί να υπάρχει μια παρέκκληση συν μείον τρία. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμά το ελεγκτικό συνέδριο. Παίρνουμε χιλιάδες περιπτώσεις και τις εξετάζουμε. Καταλήγουμε σε μια στατιστική. Η στατιστική αυτή αντανακλά βάσει μαθηματικών στατιστικών μεθόδων με κάποια αληθοφάνεια, με κάποια ποστά πιθανότητων, την πραγματική κατάσταση. Με τα νούμερα που χρησιμοποιούμε, τον όγκο του δείγματος που χρησιμοποιούμε, καταλήγουμε σε μία πιθανότητα 95% όσον αφορά το ποστό σφάλματος. Ε, ε, και συν Όταν λέμε 2,4% είναι το ποστό σφάλματος, μπορούμε να πούμε με μία πιθανότητα της τάξης του 95% ότι το πραγματικό ε, ποσοστό σφάλματος ε, κινείται μεταξύ 2,3 και 2,4. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο, γιατί βεβαίως ε, στηριζόμαστε σε μία πιθανότητα, έστω και αν είναι μία πιθανότητα 95%. Λοιπόν, γι' αυτό προσπαθούμε σε ορισμένους ε, τομείς να μην ε, δημοσιοποιούμε τα αποτελέσματα όταν ε, δεν έχει κανένα νόημα από στατιστική άποψη. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όταν κινούμεθα με ποστά σφαλμάτων. Το σύστημα αυτό προσκρούει αυτόματα στα όρια του. Όσο περισσότερο βελτιώνεται το ποστό σφάλματος, τόσο ε, μικρότερη είναι η αξιοπιστία ε, σε λεπτομέρειες. Αλλά ε, δεν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε εδώ ακριβείς μετρήσεις όσο να αφορά αυτό το οποίο είπε η κυρία Σμιτ. Δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω διαβάσει αυτό που δημοσιεύτηκε. Ξέρω ότι μόνο χτες έγινε μία συνέντευξη τύπου ε, στις ε, Βρυξέλλες, όπου το παρουσιάσαμε την έκθεση, αλλά με τον όρο ο τύπος να μην δημοσιεύσει την έκθεση χτες. Σήμερα μπορούσαν να το δημοσιεύσουν. Ε, βεβαίως έγιναν κάποιες επιμέρους ε, συζητήσεις με τους συναδέλφους αλλά βάσει της ίδιας ε, βασικής αρχής, να μην δημοσιοποιηθεί η έκθεση δηλαδή. Και τη διαδικασία αυτή την ε, συμφωνήσαμε γιατί σήμερα είμαστε στο Στρασβούργο, οι ανταποκριτές μας είναι στις Βρυξέλλες ε, δεν μπορούσαμε να δώσουμε ταυτόχρονα, δεν μπορούσα να δώσω ταυτόχρονα δύο συνέντευξεις τύπου. Εγώ βεβαίως από τη δική μου πλευρά θα δω ακριβώς ε, τι έχει γίνει. Τώρα, όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια, εγώ πριν, όταν εξελέγην πριν από τρία χρόνια πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ασχολήθηκα με το θέμα αυτό της αναπτυξικής βοήθειας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το εξή. Θα πρέπει πάντα να δούμε τι γίνεται μεταξύ των επιδόσεων από τη μία πλευρά και από τη συμβατότητα από την άλλη. Ε, εδώ υπάρχει ένα πεδίο δυνάμεων και ε, το ίδιο ισχύει για την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι μια διαδικασία με μικρό ποσοστό σφαλμάτων. Γιατί πληρώνω ε, και όταν τα χρήματα φτάσουν στην σωστή υπηρεσία δεν υπάρχει ποστό σφάλματος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά τα χρήματα. Άρα χρειάζεται εδώ μια εντατική και συστηματική διαδικασία παρακολούθησης. Γιατί ε, πολλές φορές και αν δεν υπάρχει αυτή η διαδικασία παρακολούθησης τελικά δεν ε, εκπληρώνεται ο ευκταίος ε, στόχος. Ε, υπάρχει όπως σας είπα ένα πεδίο ε, αντικείμενων, αντικρώμενων ε, δυνάμεων εδώ, ένας σχετισμός μεταξύ όλων αυτών των όρων. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία ανάθεσης έργων, όπως είπε ο κ. Τσέλερ, είναι μια απόδειξη ότι ότι όσο πιο πολύπλοκο, όσο αυξάνεται ο βαθμός πολυπλοκότητας σχέση με τις ρυθμίσεις, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των σφαλμάτων. Και εάν υπάρξει μια απλούστευση στη διαδικασία ανάθεσης, τότε θα μειωθεί και το ποσοστό σφαλμάτων. Αναφερθήκατε στο, στα, γρήγορα, στα τρένα μεγάλης ταχύτητας. Πράγματι, εδώ θα πρέπει να γίνουν πιο διεξοδικές έρευνες και θα πρέπει να εκπονηθεί ε, μια σχετικά έκθεση που αφορά ακριβώς ε, αυτά τα τρένα αλλά ε, υψηλής ταχύτητας αλλά διασυνοριακά. Όσα είπε ο κύριος Μπάλερτ θα ήθελα να πω το εξή. Το ελεκτικό συνέδριο δεν επιλέγει τα μέλη του τα μέλη προτείνονται από τις χώρες μέλη και οι χώρες μέλη στο... Ε, έχουν εντελώς διαφορετικές παραδόσεις σε σχέση με το πώς ορίζουν τα μέλη τους. Ε, και αυτές οι εθνικές παραδόσεις γίνονται σεβαστές ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά τι δικέ μα δαπάνε, τα δαπάνε του δικού μα προπολογισμού, μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι όλε μα οι δαπάνε εγκρίνονται από την αρχή του προπολογισμού και κατά τα άλλα, εμεί ω εξωτερικό. Ε, έχουμε και ένα εξωτερικό ελεγκτή που μας ελέγχει Αυτά. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Επίτροπος. Κυρία Πρόεδρε, μετά από τις ε, περιεκτικές ε, διευκρινήσεις του κυρίου Λαζάρου και του κυρίου Λένε, θα περιστώ στα εξή. Η έλεγχή μας είναι εξάντε από τη μία, εξπόστα από την άλλη. Και είναι ε, ξεκάθαρα το εξή. Πριν από την υλοποίηση του προγράμματο και τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματο. Ε, κάνουμε κάποιες διαπιστώσει, αλλά δεν καλύπτουμε όλο το φάσμα των πιθανών ε, διαπιστώσεων. Οι, αυτές που γίνονται εκ των υστέρων ε, διαλευκάνουν εκ των υστέρων μια διαδικασία και την υλοποίηση ενός προγράμματος. Άρα είναι απολύτως φυσιολογικό με αυτή τον έλεγχο εκ των υστέρων να προβούμε σε κάποιες ε, διαπιστώσεις και ε, με τον τρόπο αυτό το ποσοστό σφαλμάτων μειώνεται, γιατί κάνουμε κάποιες διορθώσεις. Ε, έγινε η κριτική ότι δεν υπάρχουν ποσοστά όσον αφορά τις χώρες μέλη. Πράγματι, στη συνοχή γίνονται, καταμερίζονται κάποια κονδύλια αναχώρα ή αναπεριφέρεια. Το πρόγραμμα Juncker, το Ταμείο Juncker δεν εξετάζει χώρες οι, οι περιφέρειες, αλλά εξετάζει την καταλληλότητα ενός προγράμματος ε, και την, ε, το κατά πόσο είναι υλοποιήσιμο. Υπάρχουν χώρες και περιφέρειες όπου τα μερίδια δεν είναι συγκρίσιμα. Υπάρχουν ορισμένες χώρες και ορισμένες ε, περιφέρειες που αξιοποιούν αυτά τα, αυτές τις δυνατότητες, άλλες όχι. Εγώ ίδιος πήγα στις, ε, απευθύνθηκα στις υπηρεσίες της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΟΗΕ για να δούμε, αν εξετάσουμε το μέλλον, ε, το, τις δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας, ιδιαίτερα όσον αφορά την Αφρική. Ε, το, στο επόμενο πλαίσιο του προπολογισμού, το, το διαμοιρασμό των κονδυλίων και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση των κονδυλίων. ξέρετε ότι η Αφρική μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Πιστεύουμε ότι τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα ε, έχουν μεγάλη εμπειρία και είναι αξιόπιστες. Και γι' αυτό θέλουμε πριν ε, διευρύνουμε το εύρος των υπηρεσιών μας να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες. Τώρα όσον αφορά την ερατότητα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης παράλληλα με τα Ηνωμένα Έθνη ή την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα και νομίζω ότι θα μπορέσουμε πολύ σύντομα να λογοδοτήσουμε ενώπιόν σας. Ε, η συγγήτρια έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι μόνο τα δύο θεσμικά όργανα, το Ελεγκτικό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και όλους τους συναδέλφους για τα χρήσιμα σχόλια που έκαναν. Ε, με εξαίρεση έναν, αλλά μια και αποχώρησε, ε, δεν θα σταθώ σε αυτόν. Είναι η δεύτερη διαδικασία απαλλαγή. Ε, γι' αυτό θα έπρεπε να σιωπά και να παρακολουθεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Όλαφ ανακάλυψε ένα μεγάλο σκάνδαλο και κατάχρηση για το ΦΥΠΙΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο και όταν αποχωρήσουν θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος ε, Μπούλοκ δεν θέλει να το ακούσει αυτό. Σε σχέση με την διαδικασία απαλλαγής, νομίζω ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Βεβαίως το ποσοστό σφάλματος έχει παγιωθεί προς τα κάτω και άρα δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Θα πρέπει όμως να μας ανησυχήσουν φαινόμενα που αφορούν τη γενική διαχείριση και την προετοιμασία του επόμενου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου σε σχέση με την διαχείριση των ΡΑΛ ως μέσων που είχε λόγο ύπαρξης αλλά τη στιγμή που ε, παγιοποιήθηκαν τα υπόλοιπα αυτά προς εκαθάριση μας δημιουργούν άλλα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, στο επόμενο πολιετές η Επιτροπή και το μέσον Invest Europe θα προσπαθήσουν να κατανείμουν καλύτερα τον κίνδυνο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που, μας, ε, που με απασχολεί, στο οποίο αναφέρθηκε ο συνάδελφος ε, Πυρίνσκι. Δηλαδή να δούμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά δημιουργούμε έτσι μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ κρατών και περιφερειών και μεταξύ πολιτών θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό. Ο κύριος Τιγκερ είπε πολύ σωστά ότι θα πρέπει να δούμε το ποσοστό σφάλματος αναχώρα. Θα δούμε λοιπόν που γίνονται και οι μεγαλύτερες ε, καταχρήσεις στις οποίες αναφερθήκαμε. Γιατί ε, άλλοι έχουν τη φήμη και άλλοι προχωρούν στο έργο. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να έχουμε μία ιεράρχηση στις χώρες, ως προς τις χώρες, πρώτη, δεύτερη και τρίτη κατηγορία. Και αυτό θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε, γιατί όπως είπε και ο Μπόκουσλαβ, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία ήταν ένα συνεκτικό στοιχείο για να μειωθούν οι ανισότητες εντός και εκτός οίκου. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το μάθημα στο όνομα της ε, διαφάνειας αποκλειστικά. Γιατί ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι για τους λαϊκιστές. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και η Επιτροπή στην επόμενη Ολομέλεια θα υποβάλει την ε, έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λένε και τον κύριο Λαζάρου που μας άνοιξαν τις πόρτες γιατί μαθαίνουμε πολλά από εσάς για να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε και εμείς τις αντιδράσεις μας σε αυτή την έκθεση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την γραμματεία γιατί εγώ ευεργετούμε από τη δική σας πείρα. Ελπίζω να φτάσουμε σε ένα αίσιο πέρα στα πλαίσια της διαδικασίας απαλλαγής. Θα ήθελα και εγώ να σας ε, ευχαριστήσω. Τώρα ήρθαμε στο τέλος του σημείου 5 της ημέρης διάταξης. Για το 6 δεν έχουμε τίποτα η επόμενη συνεδρίαση είναι Τετάρτη στις 9 το πρωί με ένα workshop για την ε, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εργασίας μας και μια βελτίωση της επικοινωνίας. Ε, στις 11 έχουμε ψηφοφορίες. Ευχαριστώ πολύ. Πέρας της ε, συνεδρίασης.